Uh, ladies and gentlemen, if you could uh, please take your seats and uh, we... Ο πρόεδρος, καθίστε σας παρακαλώ να αρχίσουμε. Θα προεδρεύσω εγώ, κατέδυση του πρόεδρου μας που είναι σήμερα απόν. Έχω ορισμένες ανακοινώσεις καθώς και άλλα θέματα τα οποία θα ήθελα πρώτα να θέσω υπόψη σας και πρώτα σε σχέση με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως και πριν σας ζητήσω επισήμως να την εγκρίνετε, έχω δύο-τρεις αλλαγές να θέσω υπόψη σας, στο χρονοδιάγραμμά μας δηλαδή, και σας τα λέω, στο τρία αγώνας κατά των απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της, Ένω, της Ένωσης με χρήση του ποινικού δικαίου. Αυτό θα αρχίσει στις 11, αντί να αρχίσει πριν από 8 λεπτά βέβαια. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή που μάλλον θα την προσέξατε ήδη. Στο υπαριθμόν 4 δια, διαδικαστικές ε, για παιδιά που μπαίνουν σε ποινικέ διαδικασίες και για ε, υπηκόους τρίτων χωρών για εθελοντικές υπηρεσίες και ΟΠΕΡ κλπ. Όλα αυτά είναι, θα συζητηθούν για τι διαπραγματεύσει για τον τριμερή διάλογο. Αυτό, αυτό λοιπόν το θέμα το μεγάλο σήμερα αναβάλλεται. Το υπαριθμόν 10 τώρα, σχέδιο τροπολογίας υπαριθμών, τροποποίησης υπαριθμών 5 στο γενικό προϋπολογισμό του 2015 και αυτό αναγκαζόμαστε δυστυχώ να το αναβάλουμε. Το υπαριθμόν 7 που είναι η εξουσιοδότηση της μέλη να κυρώσουν το πρωτόκολλο του 2014 για την Forced Labor Convention του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και για θέματα που έχουν σχέση με το ποινικό δίκαιο θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα στις 3.30 αντί στις 4. Ένα νέο θέμα, 11.1, ο οργανισμός δηλαδή θεμελιωδών δικαιωμάτων και η έκθεσή του για την βαριά εκμετάλλευση εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα. Νέο θέμα 11.2. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για τον εντοπισμό και απόσυρση επιγραμμικού εξτρεμιστικού υλικού του κ. Ντεπρέ θα συζητηθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα. Και αν δεν έχετε ιεσδήποτε ενστάσεις, τότε θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Ε, μπορώ να θεωρήσω λοιπόν ότι την εγκρίνεται. Ε, τώρα έχω και ορισμένε ανακοινώσει. Και πρώτα, σας ενημερώνω ότι το καθεστώς διερμηνίας σήμερα δεν προβλέπει δανέζικα, λετονικά, κροατικά και, και τα Ιρλανδικά, τα κελτικά αν θέλετε. Αυτό ελπίζω να μην σας δυσκολεύσει. Δεύτερο, η αποδοχή των συστάσεων των συντονιστών υπό την ισχύ του άρθρου 205 και πρώτα διορισμός εισηγητού γνωμοδοτήσεως. Ο κύριος Νίντερ Μούλερ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το σχέδιο τροποποίησης παριθμών 5 του Γενικού Προϋπολογισμού 2015. Εκεί αρμοδία επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρόκειται για γνωμοδότηση όπως ε, προανέφερα Επίσης τώρα οι ρυθμίσεις για τις εργασίες μας, έγκριση προτάσεως ψηφίσματος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια. Συμφώνησαν σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και στη χρήση μόνο της αγγλικής ως γλώσσης εργασίας ή συντονιστές. Οι πολιτικοί σύμβουλοι δηλαδή και η Γραμματεία θα συνεργαστούν στο τεχνικό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμβιβασμού. Σε δεύτερο, χρονοδιάγραμμα και διαδικασία για τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για τον προπολισμό του 2016. Έτσι είναι. Εδώ συμφώνησαν οι συντονιστέ επί τη 25 η Αυγούστου 6 το απόγευμα ω προθεσμίες καταθέσει τροπολογιών και θα δουλέψουν μόνο στα αγγλικά. Επίση, ε, δικαστικέ αποφάσει για πράξεις του πρώην τρίτου πυλώνα και για τις υποθέσεις c 317 κάθος 13, C 679 κάθος 13 και c 540 κάθος 13 και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας θα γράψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσει να υποβληθεί ένα πρόγραμμα εργασιών για την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας των μέτρων αυτών. Τώρα, το αστικό δίκαιο για την ρομποτική ομάδα εργασίας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θεωρούμε, θεώρησαν μάλλον οι συντονιστές, ότι θα πρέπει η Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών να αντιπροσωπεύεται. Ο πρόεδρος θα γράψει στον πρόεδρο της Νομικής Επιτροπής και όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν. Επίσης υπάρχουν και έξτρα συνεδριάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και προβλέπονται στις εξή ημερομηνίε. 5η 4η Ιουνίου το απόγευμα. Δευτέρα 8η Έκτου στο Στρασβούργο. φαντάζομαι ότι είναι η συνηθισμένη ε, κατά τις 7. Επίσης την 5η, 25η έκτου, πάλι το απόγευμα. Να προχωρήσω τώρα ταχαίως στα ψηφίσματα του άρθρου 133 του κανονισμού. Οι συντονιστές θεωρούν ότι δεν απαιτείται follow-up για τα εξή ψηφίσματα, για τις εξή προτάσεις ψηφισμάτων. Και πρώτα, του κυρίου Πατριτσέλο για την βελτίωση της νομοθεσίας 604 πάλι του κυρίου Πατριτσέλο για διεθνείς ε, για την διεθνή απάτη και την χρηματοδότηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας των κυρίων Σαλβίνη και Μπιζότο για την cyber security του κυρίου Καπούτο για text και data mining και copyright πάλι Καπούτο για την ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας του κ. Πατριτσέλο για τις αιτήσει πολιτικού ασύλου σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Μπιζότο. Για το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων από την Αφρική. Μπιζότο. Για την ηλεκτρονική υγεία. Πατριτσέλο. Για την έλλειψη κοινού ορισμού τρομοκρατίας στις χώρες μέλη. Πάλι Πατριτσέλο. Για τον αγώνα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας. Πάλι Πατριτσέλο. Εδώ τι λέει που είναι στα γαλλικά. Α, μάλιστα, διεθνής, διεθνής μάλλον συντονισμός διεθνών εκδηλώσεων, πάλι ο πολυγραφότατος Πατριτσέλο, για την ανάπτυξη μέτρων για την παροχή ε, ενίσχυσης σε ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι, πάλι Πατριτσέλο, και τέλος για την αναστολή της ισχύω συμφωνιών του Σέγγεν Αρναούτου. Τώρα, αναφορές. Άρθρο 126 του κανονισμού. Οι συντονιστές θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να δοθεί συνέχεια στην υπαριθμό 1073 κάθετος 14 Χόρχε Πίτα Πέρες για την βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, συμφώνησαν οι συντονιστέ να αποστείλουν γνωμοδότηση υπό τη μορφή επιστολή για την αναφορά 063-14 του Σβέν Μούλερ, Γερμανού, για θέματα τελών που εισπράττουν οι Αμερικανικές αρχές για την έκδοση προξενικών θεωρήσεων. Αυτό θα κυκλοφορήσει μεταξύ των συντονιστών. Τώρα κατάλαβα γιατί ο πρόεδρος μου ανέθεσε να διευθύνω τη σημερινή συζήτηση. Δέχεστε αυτές τις συστάσεις των συντονιστών. Υπό την ισχύ του άρθρου 205. Αν δεν ακούσω κανέναν τότε θεωρώ ότι είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ή μιλήστε τώρα ή εισηγήστε για πάντα, όπως νομίζω είπε κάποτε κάποιος με μαύρα στη γυναίκα μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για τον κύριο Τέρκ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο λοιπόν, θα πρέπει να φύγει πολύ σύντομα το πρόσωπο αυτό. Προχωρώ τώρα στην κατάσταση στην Μεσόγειο και για την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της μετανάστευσης. Η κυρία Μαρτσέλα νομίζω είναι παρούσα. Ως συνεισηγητής, νομίζω ότι υπάρχει και άλλη συνεισηγήτρια από την κυρία Κένγκη που δεν είναι παρούσα πάντως. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εφόσον συμφωνείτε κυρία Μαρτσέλα, επειδή έχουμε προσκεκλημένους που θα λάβουν το λόγο επί του θέματος, είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε μια παρουσίαση πριν λάβετε το λόγο αν συμφωνείτε. Είναι κάπως ασύνηθιστη η διαδικασία. Διότι έχουμε κοντά μας δύο ε, μάλιστα προσκεκλημένους σήμερα. Τρεις μάλιστα, τρεις. Θα παρουσιάσω τους άλλους ομιλητές σε λίγο, αλλά πρώτα χαίρομαι που μαζί μας είναι ο, Φόλκ, ο κύριος Φόλκε Τέρκ, που είναι Assistant High Commissioner για την προστασία, του Ηνωμένου Εθνών δηλαδή, των προσφύγων και θα προβεί σε παρουσίαση για το θέμα αυτό που έχουμε στην ημερησία διατάξη μας. Όπως είπα, βιάζεται να φύγει. Άρα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω θα προλάβουμε να τους πούμε λίγα πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι την συνάδελφο μου, κυρία Ματσέλο, και θα παρακαλέσω τον κύριο Τόρκ να αναλάβει αυτός ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, ότι πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τη συνεδρίασή σας. Θα πάω σε μια άλλη συνάντηση σχετική. Είναι το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράκ. Και έχει ήδη ξεκινήσει και δυστυχώς πρέπει να πάω και εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει στα θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης και ειδικότερα για την κατάσταση στη Μεσόγειο. Όπως ξέρετε από πλευράς της ΥΠΑ της Αρμοστίας παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα προσεκτικά αλλά και συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αφήξεων μέσω θαλάσσης. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, αλλά οι αριθμοί φέτος έχουν αυξηθεί. 89.000 έχουν καταγραφεί αφήξεις φέτος. Ξέρουμε ότι ε, ακόμα και στην αρχή του χρόνου δεν είναι η καλή εποχή για τέτοιου είδους μετακινήσεις, αλλά δυστυχώς βλέπετε τι αύξηση υπήρξε είναι σφαιρικό φαινόμενο, δεν είναι αποκλειστικό για τη Μεσόγειο. Εγώ προέρχομαι από ένα ταξίδι στην Παγκόγκ που έκανα και, και εκεί όπως ξέρετε συμβαίνουν αντίστοιχες ε, κινήσεις από μικτές εθνοτικές ομάδες. Βλέπουμε ότι ιδιαίτερα η Ελλάδα έχει επηρεαστεί αρνητικά μέχρι τώρα δεν υπάρχουν τόσο πολλές αφήξεις τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, ανάμεσα μάλιστα στην Τουρκία και στην Ελλάδα και αν δει κανείς τις στατιστικές είναι ξεκάθαρο ότι σχετικά με την Ελλάδα οι περισσότεροι από τους αφικνιωμένους είναι πρόσφυγες, Σύριοι περισσότεροι, αλλά και κάποιοι Ιρακινοί και γι' αυτό η συνάντηση για το Ιράκ σήμερα είναι σημαντική. Και επίσης είναι και προερχόμενοι κάποιοι πρόσφυγες από Σομαλία και Ερυθρέα. Έχουμε λοιπόν θέματα εδώ, απαιτούνται με τις χώρες αυτές όπως η Ελλάδα πολλά μέτρα αλληλεγγύης, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Γιατί βλέπουμε να συμβαίνει το φαινόμενο αυτό την παρούσα στιγμή. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Πρώτον, είδαμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κάποιες περιφερειακές συγκρούσεις να μην επιλύονται και επίσης κάποιες καταστάσεις σειράξεων οι οποίες ε, ξέσπασαν στη Λιβύη. Ιδιαίτερα μας απασχολεί πολύ και μας ανησυχεί η Λιβύη σε διάφορα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η Λιβύη στην παρούσα στιγμή δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει να λαμβάνει κάποια μέτρα συνοριακού ελέγχου και ανταπόκριση σε θέματα μεταναστευτικά ρεύματα και σε θέματα ασφάλειας και στο εσωτερικό της χώρας δυσλειτουργεί θα έλεγα η διακυβέρνηση της χώρας αυτής. Έχουμε και την συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Συρία Ακόμα και τώρα πολλοί φεύγουν από τις μάχες. Είναι ο πέμπτος χρόνος που διαρκεί η σύγκρουση αυτή και έχει αρχίσει να επικρατεί ε, στα πλαίσια των ε, μαζικών μεταναστευτικών πληθυσμών της Συρίας. Ξέρετε ότι έχουν πάει στο Λίβανο 1.200.000 Σύριοι, παρότι η χώρα έχει 3,5 εκατομμύρια και 600.000 στην Ιορδανία, 1.700.000 στην Τουρκία. Μιλάμε για τρομακτικούς αριθμούς στις γειτονικές χώρες και παρατείνεται η σύγκρουση, παρατείνεται η υποχρεωτική μετακίνηση και κάποιοι χάνουν την ελπίδα τους στην αποκατάσταση της ε, χώρας τους και προσπαθούν να ξεφύγουν επιλέγοντας την μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση. Αυτές οι καταστάσεις ε, βέβαια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, ε, μεμονωμένα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση γενικότερα για τα θέματα της μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Η εμπειρία μας μπορεί να είναι χρήσιμη ε, σίγουρα και κάποια μέτρα εσωτερικής αλληλεγγύης, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή 40.000 προσφύγων σε, από τέσσερις ε, χώρες, κυρίως από Ιταλία και Ελλάδα, είναι ένα καλό μήνυμα θα έλεγα αλληλεγγύης προς τις χώρες οι οποίες έχουν πρώτε στη και υπάρχει επίσης και ε, θέμα ανάληψης ευθύνης πλέον για την κατάσταση. Ένα άλλο σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την επανεγκατάσταση. Οι συζητήσεις που κάνετε είναι να βρεθούν και άλλες νομικές εναλλακτικέ λύσεις. Φυσικά και εμείς συμμετέχουμε, εμπλεκόμεθα στην προσπάθεια της ε, επανεγκατάστασης. Ε, πέρυσι είχαμε, διαχειριστήκαμε 80.000 ε, παλινοστούντες με διάφορους τρόπους και σε διάφορες περιοχές. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι στην Ευρώπη πράγματι ε, ε, έχει γίνει δουλειά αλλά πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 24.000 θέσεις είναι πολύ καλή αλλά λόγω των τρομακτικών αναγκών τις οποίες αντιμετωπίζουμε έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει κατεπίγουσα ανάγκη αύξησης των αριθμών αυτών εξετάζεται εναλλακτικέ λύσεις σε επίπεδο νομικό. Εμείς έχουμε, δώσει, έχουμε εκδώσει μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτών των εναλλακτικών πρακτικών σε υπόλοιπες χώρες, στον υπόλοιπο κόσμο, το οποίο καταστήσαμε διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφερθήκαμε στα θέματα, ας πούμε, ανθρωπιστικής εισδοχής, Είδαμε ότι η Γερμανία είναι πρωτοπόρος προς την κατεύθυνση αυτή σε σχέση με τους ήρου. όπως επίσης και ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης δαπανών, private sponsorship programs, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, θέματα κοινωνίας των πολιτών, ε, ομολογίες, οργανώσεις θρησκευτικέ, ανθρωπιστικές θεωρήσεις ε, που ισχύουν σε χώρες όπως η Βραζιλία ε, εισδοχή, αποδοχή εισδοχής ε, συγγενών, ε, ενοποίηση οικογενειών και εσωτερική κινητικότητα. Είναι σημαντικό να δει κανείς ότι ιδιαίτερα του Σύρους και του Ιρακινούς μήπως θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα σχήματα εργασιακής κινητικότητας που ισχύουν. Και φυσικά και το θέμα της επανεγκατάστασης είναι σημαντικό θέμα, είναι μια σημαντική νομική εναλλακτική λύση, την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην υποχρεώνονται να παίρνουν ε, πλοία τα οποία είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα λάβετε υπόψη. Περιμένουμε να μας στηρίξετε, περιμένουμε να μας βοηθήσετε ιδιαίτερα στο πλαίσιο το βορειοαφρικό και το μεσανατολικό έτσι ώστε να υπάρχουν νομικές εναλλακτικές λύσεις ε, στα πλαίσια κάποιων παραμέτρων και κριτηρίων βέβαια. Αυτά δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να παραμείνω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας κύριε Τούρκ. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Ε, ξέρω ότι έχετε ερωτήσεις. η συνάδελφος του κυρίου Τούρκ, η κυρία Κάντλα, θα παραμείνει και μπορεί ίσως ε, να μεταφέρει τις ερωτήσεις σας. Θα δώσω το λόγο τώρα μετά από τον κύριο Τούρκ και αφού ακούσουμε τους συνεισηγητές θα δώσουμε σε άλλους δύο ομιλητές το λόγο, έκτακτους. Είναι λίγο εκτός συνηθίων μας αυτή η διάταξη, αλλά είναι αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Τούρκ, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Θα επιστρέψω τώρα στην ημερήσια διάταξη και όπως είπα η συζήτηση αυτή αφορά την κατάσταση στην Μεσόγειο και την συνολική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα μετανάστευσης. Μέτσολα και Κιάνγκε είναι οι συνεισηγήτριες. Η κυρία Κιάνγκε θα έρθει λίγο αργότερα σήμερα. Είναι δύο θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν σήμερα. Καταρχάς η ανάπτυξη και η χάραξη ασφαλών οδών και δρομολογίων για τους ε, πρόσφυγες και τα θέματα της ουσιαστικής ε, εφαρμογής ε, των ρυθμίσεων που ισχύουν διεθνώς και τον ρόλο της ΙΑΣΟ. Θα ζητήσω κυρίως από την κυρία Μέτσολα σαν συνεισηγήτρια να μας ε, κάνει τη δική της παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα. and the migration Πολλή συζήτηση γίνεται για το θέμα της μετανάστευσης, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, και όσοι αναζητούν προστασία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά λέω ότι χανόμαστε στα στατιστικά στοιχεία όταν μιλάμε για μετανάστευση και ίσως είναι πολύ εύκολο να ξεχνάμε κάθε φορά που σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας και το γεγονός ότι πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει και μια ζωή και μια ανθρώπινη ιστορία. Αυτό το έχουμε ξαναδεί και ξαναδεί μετά από κάθε τραγωδία στις ακτές των χωρών μας ότι το ξεχνάει ο κόσμος μέχρι την επόμενη φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερους πνιγμούς στη Μεσόγειο που και διαπιστώνουμε τότε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτε για να λύσουμε το πρόβλημα, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα. Η νομοθεσία, ξέρετε, δεν μπορεί να δημιουργείται εν κενό. Εμεί ω νομοθέτε πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε τι οδηγεί τον κόσμο στη φυγή, τι εμπόδια αντιμετωπίζει και πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα και σε επίπεδο κράτων μελών μπορεί να βοηθήσει για την αντιμετώπιση των εμποδιών αυτών. Αν δεν έχουμε μια ολιστική ε, προσέγγιση που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, θα καταλήξουμε πουθενά. Μια από τις πτυχές είναι να δούμε ασφαλείς ε, και νόμιμες οδούς ε, για όσους αναζητούν προστασία υπάρχουν, ποιε είναι αυτέ οι οδοί και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα πριν πέσουν στα χέρια διακινητών ή ανεβούν σε σαπιοκάραβα και κινδυνεύσουν να χάσουν τη ζωή του στη θάλασσα. Έχουμε και το φρούριο Ευρώπη βέβαια που δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, και η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αλλά μια πραγματικότητα που πρέπει να τη διαχειριστούμε, όπως είπε και κάποιος. Ε, και σίγουρα χρειάζονται ασφαλείς διόδι για όσους χρειάζονται προστασία. Αυτό πρέπει να ενταχθεί ως αναπόσπαστο τμήμα ενός συστήματος πρέπει να αποφύγουμε τη διακίνηση και την ε, διακίνδυνευση ζών. Η Επίτροπος ε, ε, Μέλστρομ είχε πει ότι η παροχή ασύλου ή η αίτηση ασύλου ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα λαχείο ή ένας λαχνός. Και είχε δίκιο. Υπάρχουν ανθρωπιστικοί λόγοι που μας κάνουν να πρέπει να λάβουμε μέτρα. Έχουμε τη μετεγκατάσταση ως επιλογή. Κάθε κρατοσμένος πρέπει να παίξει το ρόλο του και αυτό πρέπει να γίνει από κοινού από τα κράτη, αν θέλουμε να έχει ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Καλές προτάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να συμπληρωθούν και με καλές πρακτικές εφαρμογής. Η μετανακατάσταση δεν αρκεί. Πρέπει στα άτομα αυτά να τους δώσουμε εργαλεία για να μπορέσουν να χτίσουν το μέλλον τους. Έχουμε εργαλεία όπως ε, τη θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους γιατί θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα ε, να μπορεί να ισχύει αυτή η παροχή της βίζας αυτής ε, σε τρίτες χώρες και πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα υποστήριξης για μεγαλύτερη για να μπορεί να καλύψει περισσότερα άτομα αυτή η διαδικασία. Επίσης, οι εκπαιδευτικές θεωρήσεις ή η διευκόλυνση εισόδου για νέους, για να έρθουν να σπουδάσουν, να ε, εκπαιδευτούν για εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε χώρου τη επαγγελματική κατάρτιση και τη ανώτατη εκπαίδευση για του νέου μετανάστε. Επίση, η κινητικότητα ε, και η βιώσιμη ανάπτυξη θα ωφεληθούν από αυτό. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε έστω και λίγο τις χώρες να ξανασηκωθούν, ε, ξανασηκωθούν ε, στα πόδια τους χωρίς να έχουμε φυγή εγκεφάλων. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και μέτρα όπως είναι η οδηγία προσωρινής προστασίας, για παράδειγμα. Και ποτέ να μην ακούμε πια επιχειρήματα για τις μαζικές, τις μαζικές εισρωές και τι προκαλούν. Και δεν τα λέω στον αέρα αυτά. Τα βλέπουμε όταν έχουμε μια μαζική εισρωή για ένα κράτος, ε, αυτό είναι μαζική εισρωή για την Ένωση. Και σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε πότε χρειάζεται στοχευμένη βοήθεια ένα κράτος μέλος. Ό,τι αφορά το κοινό σύστημα παροχή ασύλου. Σίγουρα υπάρχει κοινή ευθύνη των κρατών μελών για υποδοχή των άσυλων με τρόπο αξιοπρεπή. Να του αντιμετωπίζουν ε, με δίκαιο τρόπο. Να υπάρχουν ε, ομοιόμορφα πρότυπα, ώστε οπουδήποτε κάνει την αίτησή του ε, το άτομο αυτό να έχει την ίδια περίπου έκβαση αυτή η αίτηση. Γι' αυτό και πρέπει το CIS να εφαρμοστεί, ε, δηλαδή το, σύστημα, δηλαδή, ε, το κοινό σύστημα ασύλου. Και το γρηγορότερο δυνατό, έγκαιρα, πρέπει να μεταφραστεί η νέα δέσμη μέτρων για το άσυλο από τα κράτη-μέλη. Στηρίζω μια καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών και την ενίσχυση της δυνατότητας άσο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής για, την για τον εναρμονισμένο χειρισμό και αντιμετώπιση κάποιων περιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ετοιμότητα και σχεδιασμό για να μπορούν και τα κράτη-μέλη να μπορούν να προετοιμάζονται εκ των προτέρων. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Δουβλίνο παραδόξως δεν θα αυξήσει τις πιέσεις στα κράτη-μέλη που πρέπει να του συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ένα υποχρεωτικό σύστημα με την κατάσταση εντός της Ένωσης. Περιμένω να δω αυτό το πρόγραμμα ή αυτή την πρόταση από την Κομισιόν αργότερα φέτος και ελπίζω να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και να εξασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών. Προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση. Θα δώσω τώρα δυνατότητα και στους δύο ακόμη ομιλητές που έχουμε στο πάνελ αλλά και στους συναδέλφου μου να πάρουν το λόγο, να συμπληρώσουν αυτά που είπα Έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο ε, της, κυρίας, ε, της κυρίας και της δικής μου έκθεσης που μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαϊτσόλα. Όμως η συνεισηγήτριά σας δεν έχει φτάσει ακόμα, κυρία Κέγγι. Οπότε προτείνω να ξεκινήσουμε τον κατάλογο των ομιλητών και τους σκιώδεις εισηγητές καταρχάς, αλλά και κάποιοι άλλοι νομίζω που σήκωσαν τις καρτέλες τους, άρα και άλλοι συνάδελφοι θέλουν τον λόγο. Θα σας παρακαλέσω όμως όλους να δείξετε κάποια υπομονή. Σίγουρα θα μιλήσετε, αλλά λίγο πιο μετά. Ναι, ναι, σας έχουμε σημειώσει και σας. Όμως, προς το παρόν κύριε και κύριοι, να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, αφού τους καλωσορίσω. Καταρχάς τον ε, δόκτορα Τίλεμαν, Associate Professor Πολιτικών Επιστημών Δημοσίων Πολιτικών Διευθυντή της ε, Μονάδας ε, Μελετών για τη Μετανάστευση στο London School of Economics και στο τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Government and European Institute. Έχουμε επίσης τον Chris Pollett, Senior Legal and Policy Officer από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξόριστων. Επίσης έχουμε τον κύριο Πασκάλ Μπρίς. Όχι. Α, θα τον είχαμε. Δεν θα τον έχουμε. Διότι έχει πάρα πολλές ανηλυμένες υποχρεώσεις και επειδή στη Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα, δεν μπορούσε να έρθει ο κύριος Μπρίς. Έχει άλλες προτεραιότητες φοβούμε για σήμερα. Οπότε, να δώσω καταρχά το λόγο στον καθηγητή Τίλεμανς, Τίλεμαν, συγγνώμη. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιες ποσοστώσεις ε, ή κάποιες κλίδες διανομής ποσοστώσεων για τους ετούντες ε, διεθνούς προστασίας, δικαιούχους και μάλιστα τρία διαφορετικά είναι αυτά τα κλειδιά διανομής που έχουν αναπτυχθεί στην θεωρία και στην πράξη. Έχετε το λόγο για να μας τα θέσετε όλα αυτά. Είναι χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω στην ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μου ζητήθηκε να εξετάσω κυρίως μία βασική πλευρά των πρόσφατων προτάσεων για τα θέματα της επανεγκατάστασης και της εσωτερικής μετακίνησης. Νομίζω ότι είναι κάποιες κλίδες αυτές που μπορεί να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε εν μέρος το πρόβλημα της κατανομής ευθυνών σε επίπεδο κρατών μελών και να προωθήσουμε το θέμα της αποτελεσματικής προστασίας των προσφύγων. Έχω την εντύπωση ότι μια Ευρώπη στην οποία μοιράζονται δίκαια οι ευθυνε είναι μια Ευρώπη η οποία θα προσφέρει και περισσότερη και πιο ποιοτική προστασία στους πρόσφυγες. Νομίζω ότι οι ποσοστώσεις και οι κλίδες κατανομής μπορεί να συνεισφέρουν πολλά. Όλοι γνωρίζουμε και το είπε ο κ. Τούρκ ότι υπάρχουν βασικές αδυναμίες στο υπάρχον σύστημα και σε σχέση με την επανεγκατάσταση, όπου πολύ λίγα κράτη-μέλη δυστυχώς συμμετέχουν, με πολύ μικρούς αριθμούς. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχει πολύ υψηλός αριθμός, ποσοστιαία, σε σχέση με τις αιτήσει που λαμβάνουμε σε αιτήσια βάση. Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ένα άλμα θα έλεγα. και πράγματι υπάρχει μια δυνατότητα, μια προοπτική βελτίωση των ισχυουσών, των ισχυουσών καταστάσεων. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει σωστή ε, κατανομή των ευθυνών. Το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Και θα ήθελα και οι υπόλοιπε χώρες να δουν τις τελευταίες προτάσεις υπό το φως των προηγούμενων εμπειριών που είχαν με ε, τους δείκτες και τις κλίδες κατανομής και σε επίπεδο κρατικό και σε επίπεδο ερευνητικό, επιστημονικό αν θέλετε, Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και τις δυνατότητες βελτίωσης των προτινομένων μέτρων. Σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής ευθυνών, πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο, ε, να κάνουμε μία διάκριση, να λάβουμε υπόψη δύο διαστάσεις. Καταρχάς, οι υπεύθυνοι για τις πολιτικές αποφάσεις έχουν επιλογές σε σχέση με τους λεγόμενους δεσμευτικούς αναγκαστικούς κανόνες και τους ε, εθελοντικής φύσεως κανόνες. Υπάρχει επίσης μια άλλη σημαντική διάκριση για τον αριθμό των διαστάσεων ε, που μπορεί να πάρει η βοήθεια των κρατών μελών. Όλες οι χώρες θα κληθούν να προσφέρουν με τον ίδιο τρόπο ή ο μηχανισμός ε, επιτρέπει κάποιες χώρες να προσφέρουν με έναν τρόπο και κάποιες άλλες με διαφορετικό τρόπο. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τις επιλογές αυτές τις οποίες σας προτείνω εδώ. Σαν παράδειγμα, όταν μιλάμε για έναν μονοδιάστατο μηχανισμό αναφερόμαστε στην οδηγία προσωρινής προστασίας. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και τα εθνικά συστήματα επανεγκατάστασης. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην προστασία των προσφύγων οικονομικά όπως η Ιαπωνία ενώ κάποιες άλλες υποδεχόμενες ε, ε, τους πρόσφυγες όπως κάποιες ευρωπαϊκές. Για τους δεσμευτικούς κανόνες βλέπουμε ότι στο πρώτο επίπεδο έχουμε την εμπειρία της γερμανικής κλίδας κατανομής ε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των γερμανικών Λέντερ. Είναι μια πρόταση η οποία αντικατοπτρίζει κάποιες από τις ιδέες και τις προτάσεις της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από την άλλη υπάρχει μια τέταρτη δυνατότητα αντισταθμιστικών ε, συνεισφορών Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στις προηγούμενες διαστάσεις, δηλαδή οι χώρες οι οποίες κάνουν περισσότερα σε επίπεδο επανεγκατάστασης μπορεί να αποζημιώνονται οικονομικά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα είναι μονοδιάστα του δεσμευτικού τύπου. Ε, υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα οικονομικής βοήθειας. Ε, θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Πώς μπορεί οι υπάρχοντες εθνικοί μηχανισμοί που προτάθηκαν εδώ και αρκετό καιρό ε, να συνδεθούν με αυτά τα οποία είδαμε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένοι εξημών θυμούνται ίσως. ότι κάποιες ε, πολιτικές ομάδες είχαν ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες για την πιθανότητα εφαρμογής ε, ε, του γερμανικού συστήματος ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το είχε προτείνει και η γερμανική κυβέρνηση ήδη στην αρχή της δεκαετίας του 90, αλλά δεν υποστηρίχθηκε η πρόταση αυτή τότε. Είναι όμως κάτι το οποίο ουσιαστικά μπορεί να σχηματίσει την βάση, να αποτελέσει τη βάση του συστήματος ε, με τις κλίδες που μπορεί να και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το σύστημα Königstein λοιπόν. Η πρόταση αυτή βασιζόταν σε δύο βασικά κριτήρια, σε δύο κλίδες κατανομής στο εσωτερικό του μηχανισμού. Καταρχάς οι μεμονωμένοι αιτούντες προστασία έμπαιναν σε συστήματα κατανομής σε επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη από τη μία τον τον αριθμό του πληθυσμού και από την άλλη το ΑΕΠ της κάθε περιοχής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέτουν το θέμα της επανεγκατάστασης όπως επίσης και το θέμα της εσωτερικής μετακίνησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο, ένα επιπλέον παράγον, τον οποίο δεν είχαμε στο παρελθόν, δεν είχε προταθεί στις προηγούμενες συζητήσεις. 20.000 θέσεις ε, <clears throat> θα καταστούν διαθέσιμες ε, στην επόμενη διετία. Έχουμε 40.000 δυνατότητες εσωτερικής μετακίνησης από την ε, Ελλάδα και την Ιταλία σε προσωρινή βάση. <clears throat> Και αυτό που βλέπουμε σαν αλλαγές σε επίπεδο, σε επίπεδο κλίδας κατανομής είναι ότι συνδέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια μεταξύ τους ε, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο τον αριθμό του πληθυσμού, όχι μόνο το ύψος του ΑΕΠ, αλλά και τον αριθμό των προσφύγων που έχουν ήδη αποδεχθεί και τον αριθμό των προσώπων που έχουν ήδη μετακινηθεί, όπως επίσης και τον δείκτη της ανεργίας στη χώρα υποδοχής που αποδεικνύει εν πολύ την δυνατότητα απορρόφησης. Συμπληρωματικά, αυτό το οποίο έχουμε τώρα, είναι κάποια συνοδευτικά επίσης οικονομικά μέτρα, οι χώρες υποδοχής σαν παράδειγμα και για εγκατάσταση και για μετακίνηση θα πάρουν αναπρόσωπο 6.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται ε, ε, ίσως να προσαρμοστεί στο μέλλον προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Λοιπόν, πώς τώρα οι προτάσεις αυτές συγκρίνονται με τις ισχύουσες ή με αυτές που ίσχυαν στο παρελθόν. Καταρχάς θα πρέπει να παρατηρήσουμε κάποιες, κάποια θέματα τα οποία μπορεί να τεθούν σχετικά με την πρόταση αυτή θυμίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιες βελτιώσεις. Ε, μιλάμε για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Υπάρχουν όμως και ορισμένα θέματα που πρέπει νομίζω να υπογραμμιστούν. Ένα από τα θέματα αυτά, και αυτό είναι κάτι το οποίο η κυρία Μέτσολα ήδη ανέφερε, είναι ο μηχανισμός ε, εκκίνησης εφαρμογής του συστήματος, τον οποίο ονομάζω ad hoc, δηλαδή ε, δεν είναι μηχανισμοί μακροπρόθεσμοι, είναι περισσότερο πιλωτικού προπαρασκευαστικού τύπου ε, συστήματα. Είναι μεμονωμένοι κάθε φορά μηχανισμοί για την επανεγκατάσταση και τα κριτήρια για τις προσωρινές μετακινήσεις των προσφύγων ε, φαίνεται ότι είναι κάπως αυθαίρετα και κάπως ασύνδετα μεταξύ τους. Για το ποιες σαν παράδειγμα χώρες θα εφαρμόσουν το σύστημα της εσωτερικής μετακίνησης Προτείνεται η Ιταλία και η Ελλάδα, αλλά όχι η Μάλτα σαν παράδειγμα και αυτό θα προκαλέσει συζητήσεις. Το δεύτερο θέμα το οποίο έρχεται στην επιφάνεια είναι ότι οι προτάσεις αυτές παρουσιάζουν πολλούς περιορισμούς ε, στις μετακινήσεις των ατόμων αυτών που χρησιμοποιούν τα προγράμματα αυτά, τα προγράμματα επανεγκατάστασης ή τα προγράμματα εσωτερικής μετακίνησης. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι περιορίζοντας τις επιλογές των ετούντων άσυλο σε επίπεδο χωρών μπορεί να δικαιολογηθεί για στόχους και για λόγους δικαιοσύνης και κατανομής των ευθυνών, ε, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι ε, μετακινούνται σε άλλη χώρα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι πρόσφυγες σε κάποιο συγκεκριμένο μέλος υφίστανται και υπόκεινται για πέντε χρόνια τον μηχανισμό του Δουβλίνου αν θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα. Και αυτό φαίνεται σχετικά δυσανάλογο σαν περιορισμός ε, μετακίνησης. Επίσης οι προτάσεις αυτές στην ουσία συνιστούν περιορισμένες κατεξαίρεση αποκλήσεις από το Δουβλίνο, από τη Συμφωνία Δουβλίνο. Λοιπόν, αυτό ε, ήδη έτσι κι αλλιώς μέσω του Συμφωνίας του Δουβλίνου υπάρχει α, άνηση και άδικη κατανομή ευθυνών. Και τέλος, ε, εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα ε, αναλογικής αντιμετώπισης κάποιων θεμάτων. Το θέμα της ε, οικογενειακής επανένωσης, σαν παράδειγμα, είναι θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί, λέει η πρόταση. Αλλά κάποιες άλλες προτιμήσεις που μπορούσαν να έχουν οι υποψήφοι, ε, σαν παράδειγμα λόγω γλώσσας ή λόγω πολιτισμικής εγκύτητας στις επιλογές τους, αγνοούνται πλήρως. Ε, και αποφασίζεται η χώρα υποδοχής με εντελώς αφαίρετο τρόπο. Ε, βέβαια κάποια επιπλέον στοιχεία ε, παράμετροι επιλογής θα αυξήσουν την περιπλοκότητα του συστήματος και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Και τέλος, αντίθετα και με άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι πρόσφατες προτάσεις δεν προβλέπουν μια πολυδιάστατη ε, λειτουργία του συστήματος, ένα πολυδιάστατο μηχανισμό. Όπως είπα υπάρχουν συνοδευτικά οικονομικά μέτρα, αλλά δεν επιτρέπεται ας πούμε η εμπορία ποσοστώσεων προσφύγων, όπως έχουν προτείνει ορισμένοι ερευνητές. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε μία πρόσφατη συνεισφορά στη συζήτηση αυτή, οι ακαδημαϊκοί Ράπαπορτ και Μοράγκα είπαν ότι μπορεί να υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια του νέου σχήματος ανταλλαγής ποσοστώσεων, εμπορίας ποσοστώσεων, που επιτρέπουν στις χώρες οι οποίες θέλουν να μειώσουν την ποσόστοσή τους να πληρώνουν κάποιες άλλες χώρες για να δέχονται περισσότερους and encourage participation και ένα τέτοιο σύστημα να βοηθήσει έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δισταγμοί ορισμένων κρατών μελών που είναι εναντίον της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή και τις κλίδες κατανομής. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί βέβαια μια κάποια δυσφορία, κάνει τη συζήτηση πιο δύσκολη αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέματα που εξετάζονται και είναι σημαντικά θέματα για τη συζήτηση. Θα ολοκληρώσω εδώ λέγοντας um, parliament, και um, ε, ότι το Κοινοβούλιο και η Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή θα πρέπει να τους συγχαρούμε γιατί κρατάει ψηλά το θέμα της κλίδας κατανομής Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όπως είπα στις δυνατότητες του συστήματος αλλά εφόσον γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνουν ένα πρώτο σκελετό αν θέλετε μέτρων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη περισσότερης δικαιοσύνης, περισσότερης αλληλεγγύης και περισσότερων ευκαιριών για τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ασφαλώς ε, θα έχουμε ερωτήσεις αργότερα εφόσον μπορείτε να παραμείνετε. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον κύριο Πόλετ που είναι εκπρόσωπος του ECRE, e, μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας 87 μη κρατικών οργανώσεων που εργάζονται ε, για να ενισχύσουν ε, μετανάστες, πρόσφυγες, εκτοπισμένους και θα ήθελα να ακούσω τώρα από τον ίδιο πού βρισκόμαστε και ποια είναι η συνέχεια που δίνεται στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Κέρκοπ, ευχαριστώ και την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών που μας προσκάλεσε στη συνάντησή σας. Μας ικανοποιεί βεβαίως πάρα πολύ η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει ως Επιτροπή ΛΥΜΕ για τη σύνταξη εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας και χαιρόμαστε επίσης για την προσοχή που χαρίζεται στο θέμα. Όπως είπε ο Πρόεδρος σας, εκπροσωπώ την ΕΚΟΕ. Όντως είμαστε μια συμμαχία 85 ε, μη κρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούμεθα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολλές μάλιστα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου και των προτύπων που έχουν εγκριθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτη. αποτελούν και βάση της εργασίας μας και βεβαίω μας απασχολούν πάρα πολύ. Έχουμε συνεργαστεί και μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν γινόταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πακέτο του ασύλου. Προσπαθούμε τώρα να παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Τα πρότυπα αυτά που αναγνωρίζουμε ότι τα πρότυπα που βρίσκονται στο κεκτημένο έχουν σημαντικά βελτιωθεί από πολλές πτυχές, βεβαίως ακόμα μας ανησυχούν ορισμένα πράγματα. Θέλουμε πάντως οπωσδήποτε να παρακολουθούμε όσο γίνεται στενότερα την εφαρμογή τους και όχι μόνο τη μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες αλλά και την πραγματική εφαρμογή τους, στην πράξη δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, καμιά φορά υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στα δύο αυτά, νομοθεσία και πράξη. Να πω λοιπόν τώρα ότι έχουμε δύο εργαλεία στη διάθεσή μας, δύο δηλαδή τράπεζες δεδομένων. Την Asylum Database που εξετάζει τις πρακτικές ασύλου, κράτησης κλπ. σε 16 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία. Έχουμε και την EDAT Database που συλλέγει νομολογία, που είναι βέβαια πολύ σημαντική ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τα δικαστήρια εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία. Γιατί σας τα εξηγώ αυτά. Όχι μόνο για να κάνω και λίγη αυτοδιαφήμιση για την οργάνωσή μας, αλλά και διότι νομίζω ότι είναι ουσιώδες όταν μιλούμε για την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, να αντιληφθούμε ότι όλες οι πτυχές, όλες οι απόψεις είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη. συλλέγεται στο ΕΑΣΟ, πολλές, λέγονται μάλλον πολλές πληροφορίες και ιδίως στατιστικού χαρακτήρα, αλλά βεβαίως και για τις ε, πρακτικές εφαρμογές και αυτό σίγουρα είναι πολύ ορθό. Αλλά πιστεύουμε ότι και η οπτική των ανθρώπων που εφαρμόζουν στην πράξη, δηλαδή των νομικών που εφαρμόζουν στην πράξη τα πράγματα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα της καταστάσεως του ασύλου στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν χαίρομαι και σας, ε, για την προσπάθεια που κάνετε και σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές τις οποίες ε, σας διαθέτουμε στη δια... μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών σας. Να σας εξηγήσω όλο τώρα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου σε 10 λεπτά βεβαίως είναι mission impossible και δεν θα προσπαθήσω καν να το κάνω. Αλλά θα προσπαθήσω να σας επισημάνω κάποια σημαντικά στοιχεία που θεωρούμε ότι παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Επί του παρόντος θα πω και λίγα λόγια για τον ειδικότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και βεβαίως του ΕΑΣΟ. Συμμεριζόμαστε την ανησυχίε που εκφράζεται στο ψήφισμά σα και που ζητείτε μια ολιστική προσέγγιση συνολική προσέγγιση δηλαδή για την χρήση, την εφαρμογή και χρήση αποτελεσματικών κοινών προτύπων. Γιατί παρόλο που έχει περάσει μια 15 ετία νομοθετικής εναρμόνισης, θεωρούμε ότι ακόμα υπάρχουν σημαντικότατες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους, αλλά και σημαντικότατες προκλήσεις και ε, για τους ε, ετούντες άσυλο να επιτύχουν σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Και ιδίως η μεγάλη ανισότητα, οι πολλές παραλλαγές, οι πολλές διαφορές στην εφαρμογή και στα νομικά πλαίσια που εφαρμόζουν οι χώρες μέλη. Και βεβαίως οι διαφορές, οι ανισότητες για τις ίδιες εθνικότητες, που εφαρμόζουν τις ίδιες εθνικότητες και η άνηση βέβαια κατανομή των υποθέσεων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά δήλωσή τη θέλει να εφαρμόσει μια κοινή προσέγγιση. Δύο λόγια μόνο για τις διαφορές στα ποσοστά αναγνωρίσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές αυτές. Γνωρίζω βέβαια ότι πίσω από του αριθμού κρύβεται μια ολόκληρη πραγματικότητα, διότι οφείλει κανεί να λάβει υπόψη και τα διαφορετικά προφίλ, διαφορέ των υποθέσεων μεταξύ του κτλ. Όμω οι ανισότητε υπάρχουν και δείχνουν ότι ακόμα υπάρχει πολύ διαφορετική αντίληψη και ανάμεσα στις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά το ποιος άνθρωπος έχει ανάγκη από διεθνή προστασία. Η ΆΣΟ βέβαια δρά, κάνει προσπάθεια για να αμβληνθούν αυτές οι διαφορές, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ε, θεμελιώδες για το πώς εφαρμόζεται το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Δεύτερο σημαντικό θέμα από τη σκοπιά των ε, τούντων άσυλο αλλά και των NGO που εργάζονται μαζί τους είναι και το επίπεδο διαθεσιμότητας των ε, εγκαταστάσεων που ε, υποδέχονται τα πρόσωπα αυτά. Υπάρχει το πρόβλημα σε πολλές χώρες, έχουμε το πρόβλημα της Ελλάδος, είχαμε το πρόβλημα της Βουλγαρίας, λίγο παλαιότερα δηλαδή πέρσι. Έχουμε ακόμα και σε άλλες χώρες όπου δεν θα το ανέμενε κανείς σε μεγαλύτερες χώρες όπως η Γαλλία. Έχουμε πρόβλημα πρόσβασης σε καταλήματα των ετούντων άσυλων. Είναι ένα πρόβλημα δομικού χαρακτήρα, διαθωτικού χαρακτήρα. Δεν είναι μοναχά ένα πρόβλημα στις νέες χώρες μέλη, αλλά οριζόντιο. Γνωρίζουμε βέβαια και το Δικαστήριο, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζει και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της πρόσβασης σε χώρους υποδοχής όταν εξετάζει διάφορες υποθέσεις. Δεύτερη πτυχή που θέλω να επισημάνω εδώ είναι η πρόσβαση σε ποιοτική νομική υποστήριξη. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι στη σχετική οδηγία έχουν προβληθεί πολλές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ανύψωση του ποιοτικού επίπεδου για τις διαδικασίες των προσφύγων, αλλά η πρόσβαση στην νομική στήριξη, νομική υποστήριξη, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της αρχής front-loading. Οι ετούντε άσυλο σήμερα στην Ευρώπη, μάλλον οι διαδικασίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες και επομένως είναι απόλυτα αναγκαίος όρος η πρόσβαση στις ε, συμβουλές ενός επαγγελματία νομικού για τους ετούντες άσυλο. Και αυτά καθορίζονται και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μέσα από μια σειρά μέτρων, δημοσιονομικές περικοπές, ε, αντικίνητρα για δικηγόρους να ασχοληθούν με θέματα ασύλου και να υποστηρίξουν ετούντες άσυλο. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τελικά στην πράξη να γίνεται όλο και λιγότερο προσβάσιμη η παροχή νομικών συμβουλών από επαγγελματίε νομικού του το άσυλο. Και ιδίω εκεί όπου είναι και πιο αναγκαίο. Για παράδειγμα, νομική υποστήριξη στα σύνορα, σε κέντρα κρατήσεω και ούτω καθεξής. Εκεί δηλαδή όπου η νομική αυτή ε, παροχή συμβουλών είναι και πιο σημαντική. Ένα τρίτο θέμα βέβαια δεν θα μπορέσω να μην πω ορισμένα πράγματα για το Δουβλίνο εργαζόμενος για τον οργανισμό που εργάζομαι. Και τα παραδείγματα που ανέφερα έως τώρα και αυτές οι ανισότητες που διαπιστώνουμε ότι υφίσταται δείχνουν ξανά ότι τα θεμέλια του συστήματος του Δουβλίνου η υπόθεση δηλαδή ότι όλες οι χώρες μέλη μπορούν να θεωρηθούν ως ασφαλείς χώρες, ότι όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τα πρότυπα ε, ε, εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, και αυτό οφείλει να ληφθεί υπόψη. Το σύστημα του Δουβλίνου αποτελεί βεβαίω τον θεμέλιο λίθο του κοινού συστήματο ασύλου στην Ευρώπη. Άρα αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Επίση, σημειώνω το γεγονό ότι ορισμένα στοιχεία του κανονισμού του Δουβλίνου, η πραγματική βάση στην οποία βασίζεται ο κανονισμός, η ιεράρχηση δηλαδή κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία οι χώρες μέλη καθορίζονται ότι είναι υπεύθυνη χώρα μέλος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Δηλαδή συχνά παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας επισημάνω είναι το άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου. Έχουμε επισημάνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει και ένα σχεδιασμό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Και επομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προλαμβάνει κρίσει μέσα στα συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό όμω δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα και διερωτώμεθα γιατί. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμό του Δουβλίνου, έχουμε αντιμετωπίσει κατ' επανάληψη περιπτώσει, ανέφερα πριν τη Βουλγαρία, αλλά επίση και η περίπτωση τη Ιταλία και τη Ελλάδο, όπου δεν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα πράγματα έως τώρα. Και έχουμε βέβαια τώρα και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 78 παράγραφος 3 που φαίνεται ότι αυτή θα πρέπει να είναι η σωστή βάση. Και εμείς βεβαίως ε, δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως επισημαίνω ότι ισχύει μονάχα για κατεπίγουσες καταστάσεις, ενώ το 33 ε, υποτίθεται ότι βοηθεί στο να προλαμβάνονται τέτοιες κρίσεις. Πολύ σύντομα τώρα, γιατί βέβαια το χρονόμετρο προχωρεί, ε, ο ρόλος του ζήτηση αυτή νομίζω ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς. Βεβαίως, η παρακολούθηση της εφαρμογής αποτελεί καθήκον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Γνωρίζουμε όμω ότι οι πόροι τη Κομισιόν είναι περιορισμένοι. Και βεβαίω έχει αγαθές προθέσει, όπω γνωρίζουμε, να ξεκινήσει και με διαδικασίε προσφυγή λόγω παραβιάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά θα ήταν όμως η Επιτροπή σα κάπου κάπου να υπενθυμίζει στην Κομισιόν τα καθήκοντά τη. Δεύτερο, θεωρώ ότι υπάρχει και η δυνατότητα για την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών να πάει να δει επιτόπου τι γίνεται η Επιτροπή σας λοιπόν, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, μπορεί να οργανώσει και επιτόπου επισκέψεις για να δει τι γίνεται και για καλές ε, πρακτικές και για κακές πρακτικές στις χώρες της Ευρώπης. Τρίτο, έχουμε και το Ταμείο Μεταναστεύσεων, Μεταναστών κτλ. που προσφέρει πόρους σε χώρες μέλη για να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του, και είναι επίση πολύ σημαντικό να δούμε αυτά τα χρήματα πώ δαπανώνται, με ποιον τρόπο δαπανώνται. Και εκεί νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει έναν εντονότερο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Κύρκοπ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Πόλετ. Ε, θα μπορέσετε και αργότερα ενδεχομένω να απαντήσετε σε ερωτήσει. Τώρα η συνεισηγήτριά μα η κυρία Κέγγε έφτασε τελικά. Έχω και μπροστά μου τον κατάλογο των ομιλητών, τους σκιώδεις εισηγητέ. Θα ήθελα όμως ίσως να δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Κέγγε εφόσον το επιθυμεί και μετά στους υπολείπου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν υπάρχει μία λύση απέναντι σε αυτή την τραγωδία η οποία χτυπά τη Μεσόγειο. Είναι κάτι το οποίο αφορά και την κοινωνία και την ασφάλεια και τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτά τα είπε ο ίδιος ο Μπαν Κιμούν, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, στην επίσκεψη την οποία έκανε πρόσφατα στη Ρώμη είναι απελπισμένες ενέργειες, απονενοημένα διαβήματα από πλευράς αυτών που προσπαθούν να ξεφύγουν από το θάνατο και την τραγωδία. Το θέμα δεν είναι η στρατιωτικοποίηση βέβαια όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας των Συνόρων. Οι πολιτικές ε, αυτές οδηγούν τους μετανάστες να ακολουθούν ακόμα πιο επικίνδυνες οδούς και να αφήνονται στα χέρια επικίνδυνων θανατηφόρων δικτύων. Πρέπει να δούμε τι απάντηση θα δώσουμε στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Ασχοληθήκαμε με τα κατεπήγοντα μέτρα σε βραχία περίοδο, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πανανθρώπινη αξία. Δυστυχώς καμία άμεση απάντηση όσο και μακροπρόθεσμη και αν είναι δεν μπορεί να αλλάξει σε βάθος την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πολιτικές και τα μέσα που διαθέτουμε και σε επίπεδο εσωτερικής και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα πρώτο υπεύθυνο βήμα. Τα προγράμματα μετεγκατάστασης, τα προγράμματα εσωτερικής μετακίνησης, όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Οι πρόσφατες ε, συστάσεις για 20.000 θέσεις που χρήζουν διεθνούς προστασία τα επόμενα δύο χρόνια είναι ένα πρώτο και ε, μετριοπαθές βήμα, όπως επίσης και η προσπάθεια δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων. Η διαδικασία όμως είναι μακρά η εγκατάσταση 20.000 ή επανεγκατάσταση 40.000 μέσα σε δύο χρόνια δεν θα δώσει μια εξαντλητική απάντηση στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας παρουσιάσει όπως το ζητεί το Κοινοβούλιο μια νομοθετική πρόταση. Μια πρόταση η οποία να προβλέπει έναν μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάστασης ε, με αριθμούς οι οποίοι να αντιστοιχούν στο μέτρο ενός μίας υπήρου 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Νομίζω ότι μετά από τις παρουσιάσεις σας μπήκαμε στα συγκεκριμένα θέματα της νόμιμης ε, εισόδου των ανθρώπων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, χρηστές πρακτικές, πειραματισμοί σε τοπικό επίπεδο, κάτι το οποίο μπορούμε να από το οποίο να υποφεληθούμε στο μέλλον. Πιο αποτελεσματικά συστήματα, πολύ καλύτερα από στρατιωτική αντιμετώπιση ε, του φαινομένου ή αυτών οι οποίοι παρέχουν ε, τα σκάφη με τα οποία γίνεται η είσοδος αυτή πρέπει να ασκήσουμε θα έλεγα φιλόδοξες πολιτικής και για την ολοκλήρωση των μεταναστών, την ενσωμάτωση μάλλον των μεταναστών και την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφύγων. Το, η πρόκληση μπροστά μας πρέπει να έχει σαν βασικό στόχο, είναι μάλλον μεγάλη και βασικός μας στόχος είναι η διαχείριση και ολοκλήρωση των μεταναστευτικών ραών, ραών τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ιστό των κοινωνιών που υποδέχονται αυτούς τους μετανάστες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών που, που διαχειρίζονται πρώτοι ε, την είσοδο αυτών των ανθρώπων. Σκέφτομαι στον ε, Έντσο Μπιάνκο από την Κατάνια, δήμαρχο της Κατάνιας, την Τζούζη Νικολίνη, δήμαρχο της Λαμπεντούζα και τις πρωτοβουλίες, το θάρρος και τη γενεοδορία που επέδειξαν όπως και αντίστοιχα του λαού της Σικελίας που έφτασαν μόνο την προηγούμενη εβδομάδα 15.000 πρόσφυγες. Λοιπόν, μια σωστή πολιτική ασύλου, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δουβλίνο έτσι όπως έχει σχεδιαστεί δεν λειτουργεί. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για μια σωστότερη εφαρμογή. Εμείς πρέπει να κάνουμε προτάσεις για την αλλαγή του Δουβλίνου. Κάποια νομοθετική πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν είναι σταθερή, στατική και μη μεταρρυθμίσιμη. Το 78 παράγραφος 3 της συνθήκης δείχνει ότι μπορεί να ληφθούν μέτρα τα οποία μπορεί να είναι περιορισμένα αλλά ανοίγουν τον δρόμο σε συγκεκριμένες λύσεις. Θα ήταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ε, να μην ξεχνάμε και τη συμφωνία του Σέγγεν 30 χρόνια μετά την υπογραφή του. Θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις φιλόδοξες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι χρήζουν και δικαιούνται διεθνούς προστασίας και να μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες μέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιέγγε. Και τώρα έχω έναν μακρύ κατάλογο ομιλητών. Καταρχάς όμως μία μικρή ανακοίνωση. Όσοι ανησυχείτε για τη δερμηνία προς τα σλοβακικά αλλά όχι από τα σλοβακικά. Δεν υπάρχει δερμηνία ούτε από ούτε προς. Ή αν κατάλαβα καλά, ενδεχομένω πρώτα να μιλήσετε, αλλά μην μπορείτε να ακούσετε. Αν καταλαβαίνει κανείς καλύτερα από μένα, μπορεί να μου το πει και εμένα. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στου σκιώδεις, συντονιστές και όποιον άλλο θέλει το λόγο. Δύο λεπτά ο καθένα όπως είπα, μακρύς ο κατάλογος. Οι συντονιστές και οι ισχυώδεις θα μιλήσουν για δύο λεπτά και οι υπόλοιποι ένα-ενάμιση λεπτό ο καθένας. Για να έχουμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε και τους ε, συνεισηγητές, τις συνεισηγήτρες στην προκειμένη περίπτωση και ίσως και τους ομιλητές μας. Λίγο πολύπλοκη η διαδικασία, περνώ όμως ευθύς αμέσω στην κυρία Βίξτρομ που και αυτή νομίζω πρέπει σύντομα να φύγει. Παρακαλώ έχετε το λόγο κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και κάνατε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Είμαι σκιώδη συζητήτρια της ομάδα των φιλελευθέρων. Μαζί με την Γιούντιτ Σαρτζεντίνη από την ομάδα των Πρασίνων έχουμε εκπονήσει ένα έγγραφο εργασίας ε, για τις νόμιμες ασφαλείς οδούς ε, για, την, για τους ετούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παγκόσμιων προσφύγων δεν φτάνει ποτέ στην Ευρώπη. Όσοι όμως επιθυμούν να έλθουν στην Ευρώπη, δεν έχουν και πολλές, ε, αντίθετα πολύ λίγες δυνατότητες για να φτάσουν με νόμιμο και ασφαλή τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε και τα κεκλώματα των αδίστακτων αυτών διακινητών, που είναι μια πολύ κερδοφόρα απασχόληση. Και σε αυτούς στρέφονται όσοι δεν έχουν καμία άλλη εναλλακτική. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τα θύματα στη Μεσόγειο και θέλουμε να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα, τη δράση των διακινητών και να παράσχουμε εναλλακτικές αν υπήρχαν διάβλοι ασφαλείς νόμιμοι, ο κόσμος πιστεύω είναι αρκετά έξυπνος για να, προστα... Ε, να προτιμήσει αυτές τις οδούς και όχι τις παράνομες. Υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες παροχής ε, κάποιες νομικής βοήθειας στους έτοντες ε, άσυλο, αλλά πολλές φορές είναι αντικείμενο κατάχρησης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τώρα όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο σχέδιο του δικού μας εγγράφου Αναφέρουμε κάποιες προτάσεις, ε, μιλούμε για τη μετεγκατάσταση της ε, θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, την ιατρική εξέταση, τα λεγόμενα private sponsorships επανένωση οικογενειών, ακαδημαϊκές υποτροφίες ε, και κάποια άλλα προγράμματα εργασιακής κινητικότητας. Να μιλήσω εν συντομή για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις ε, και την μετεγκατάσταση. Έχουμε το πρόγραμμα της ΥΠΑ Αρμοστίας. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα. Όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να μας ενοχλεί για να μην μπορεί να μας κάνει να ντρεπόμαστε το γεγονός ότι ενώ παίρνει... Ε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η ε, Αμερική, εμείς παίρνουμε ούτε το 12. Γύρω στα 5-6 άτομα μεταφέρθηκαν σε 15 ε, κράτη. 13 δηλαδή ε, το παίζουν πόντι πιλάτη. Σαν να μην έχουν καμία ευθύνη νύπτουν τα σχήρα τους αυτά τα 13 κράτη-μέλη. Υποχρεωτικά όμως πρέπει να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Και έτσι θα αυξηθούν και οι αριθμοί. Τώρα για τι θεωρήσει για λόγου. αυτό είναι κάτι άλλο, δεν ε, θέλω να ακρηγορήσω, αλλά και πάλι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και το κάτσο 22. Αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι να εξετάσετε τι μπορεί να γίνει με τις υφιστάμενες διατάξεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και που μου δώσατε αμέσως το λόγο για να μπορέσω να προλάβω και την πτήση μου. Uh, Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, φαντάζομαι βασιστήκατε και σε αυτά που είπε ο κύριος ε, Τίλεμαν πριν. Η κυρία Χέρς το είχε θέσει για πρώτη φορά το 2011 και μετά έχουμε την πρόταση του 2012. Ο καθηγητής αναφέρθηκε σε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν Σεσίλια. Έχουμε και τον κύριο Άλε Ο, εκ μέρους της κυρίας Στίβενς, από την ομάδα ECR. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι 20.000 λέτε για μετακατάσταση, 40.000 ε, για εσωτερική μετακίνηση. Αυτά τα νούμερα μου φαίνονται ανεδαφικά μικρά, αν τα συγκρίνουμε με το συνολικό αριθμό των ατόμων που ε, επιχειρούν ε, να εισέλθουν στην Ευρώπη, βρίσκονται σε καταβλισμού σε περιοχέ συγκρούσεων. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτά τα προγράμματα έχει, υπάρχει κάποια πιθανότητα να αποθαρρύνουν τον κόσμο από το να χρησιμοποιήσει μια παράνομη οδό. Υπάρχει τελικά λύση. Ή βολικά είναι τόσο χαμηλά αυτά τα νούμερα απλά και μόνο για να τα πλασάρουμε στους Ευρωπαίους. Επίσης ακούσαμε ότι μεγαλύτερο ε, μέρος αυτών που έρχονται στην ε, Ευρώπη δεν προέρχονται από τη Συρία ή άλλες περιοχές ε, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά οικονομικοί μετανάστες κυρίως από τη Δυτική Αφρική και αλλού. Άρα ερωτώ, η ιδέα ότι αυτά τα άτομα θα ενταχθούν στα προγράμματα εσωτερικής μετακίνησης οι αιτούντες, πρόσφυ, οι αιτούντες άσυλο κατά κάποιο τρόπο θα περάσουν από ένα ε, σύστημα διαλογής, πρώτερης διαλογής προτού μεταγκασταθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Είπε και η κυρία Μέτσολα ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, επιτυχή ένταξη των μεταναστών. Πάντως φαίνεται ότι καμία δυτική χώρα δεν κατάφερε να εντάξει επιτυχώς στους κόλπους των κοινωνιών τους τους μετανάστες που έρχονται για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι οικονομικό και κοινωνικό, αλλά και πολιτικό το πρόβλημα. Αν αυξηθούν οι αριθμοί δραματικά, πιστεύετε ότι θα μειωθούν αυτά τα προβλήματα. Πρόεδρος, όχι. Ευχαριστώ. Η Judith Sargentini είναι η επόμενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους σημερινούς ομιλητές. Η συνάδελφος Έλια Βίξτρομ αναφέρθηκε στο έγγραφο το οποίο προετοιμάσαμε και το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Να υπογραμμίσω εδώ το μνημόνιο που μας έστειλε σήμερα η ύπατη αρμοστία είναι, έχει μεγάλη εμβέλεια και είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένο έγγραφο γιατί δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην αναζήτηση νομικών τρόπων αντιμετώπισης της μετανάστευσης και προσφύγων. Το θέμα δεν είναι μόνο η κατανομή, η επανακατανομή ή η επανεγκατάσταση. Εγώ εξετίμησα δεόντως και τις επεξηγήσεις του κυρίου Τίλεμανς, αλλά να μην περιοριστούμε εδώ, νομίζοντας ότι μια τέτοια λύση θα είναι η μοναδική. Η κρίση θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση και όχι να αποστρέφουν την κεφαλή, αλλά και να συνεχιστεί φυσικά θα συνεχιστεί η προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων να έλθουν στην Ευρώπη. Ε, ας μην ε, περιοριστούμε στα της Μεσογείου. Ξέρετε ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία στην παρούσα φάση είναι δύσκολη. Στην ανατολική πλευρά πολλοί προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη ε, μέσω επίγειων οδών. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε η τουριστική βίζα και όταν οι έλεγχοι στις θεωρήσεις αυτές από τις ε, αεροπορικές εταιρείες δεν ήταν αυστηρές, τότε πολλοί ερχόντουσαν άμεσα αεροπορικά και νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους απαιτείται να επανεξεταστεί η Συμφωνία του Δουβλίνου. Έχουμε περιορίσει ε, την είσοδο στην Ευρώπη στα σύνορα των χωρών και έτσι έχουμε επιβαρύνει τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Ε, ε, θα θέσω μια ερώτηση, δεν θα καθυστερήσω άλλο. Κύριε Τίλεμαν, για την πιθανή μόχλευση, δηλαδή τι θα συμβεί εφόσον χρησιμοποιηθεί μια κλίδα κατανομής με όλες αυτές τις δυνατότητες εξαίρεσης. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει την εμπορία σε εισαγωγικά αυτών των ποσοστώσεων. Είδαμε χώρες ε, που δεν έχουν τεράστιους τέτοιους πληθυσμούς, αλλά στην ουσία ε, το θέμα είναι ποιος έκανε το αυγό η κότα ή η κότα το αυγό. Οι πρόσφυγες δεν πηγαίνουν εκεί διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ε, κίνητρα για τους μετανάστες να πάνε εκεί. Ευχαριστώ. Θα περάσω στους συντονιστές που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Σίπολ, Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα. Θα ξεκινήσω με ένα σύντομο επιχείρημα ή μάλλον με μια σύντομη δήλωση. Είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη γιατί προσπαθούμε σαν Κοινοβούλιο και Επιτροπή να αντιμετωπίσουμε το θέμα συνολικά, αλλά από ό,τι ακούμε από τις συζητήσεις και από ό,τι διαβάζουμε, τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να ακολουθήσουν την αντίληψη αυτή δεν θέλουν να καλύψουν όλους τους τομείς που οδηγούν στη μετανάστευση. Πολλές χώρες δεν θέλουν να ασχοληθούν ούτε με έναν από τους τομείς αυτούς και αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται εδώ μια κάποια ηγετική θα έλεγα στάση από πλευράς των πιο προχωρημένων στον τομέα αυτών χωρών οι οποίες πρέπει να πούν ότι πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους εμείς πήραμε τα ρίνουμε τις υπόλοιπες χώρες να κάνουν το ίδιο. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, σχετικά τώρα με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη γύρω από το θέμα της ε, προστασίας της διεθνούς με διαφορετικά επίπεδα κάθε φορά. Η εφαρμογή του νέου πακέτου ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει ανταπόκριση από πλευρά των κρατών μελών έτσι ώστε να συμμορφωθούν με αυτά τα οποία έχουν οι ίδιες αποφασίσει έτσι ώστε τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου χρόνου να υπάρξει κάποια πρόοδος. Ευχαριστώ. Την έχω βρει εδώ, ε, λόγω της Προεδρίας και γι' αυτό δεν θα πω προς το παρόν τίποτα, δεν θα πάρω το λόγο. κυρία Φεράρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τα θέματα της πρόσβασης των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη ευ... νόμιμης εισόδου αυτών των ανθρώπων σαν η μοναδική λύση στις παράνομες μετακινήσεις και σε αυτούς που εκμεταλλεύονται και εποφελούνται από την έλλειψη νομικής δυνατότητας πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα συμφωνήσω με την κυρία Κιέγκε ε, λέγοντας ότι οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές δράσεις ε, δεν θα ήταν χρήσιμες. Πιο χρήσιμο, πιο σοφό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους νόμιμους τρόπους εισόδου. Ε, δεν είμαι σίγουρη στο ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν ένα θετικό βήμα, γιατί οι προτάσεις αυτές θα καλύψουν μόνο ένα περιορισμένο αριθμό ετούν τον άσυλο και μόνο κάποιες κατεπίγουσες περιοχές, ε, καταστάσεις θα έλεγα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες νεκροί στη Μεσόγειο και δεν μπορούμε να μιλάμε για προσωρινούς μηχανισμούς. Εύχομαι το ταχύτερο δυνατόν να βρούμε κάποιους ε, μόνιμους μηχανισμούς κατανομής και συμμερισμού της ε, ευθύνης. Τροποποίηση φυσικά του κανονισμού του Δουβλίνου, το έχουν θέσει πάρα πολύ αυτό, αυτό το οποίο μου ε, προκάλεσε το ενδιαφέρον στην παρουσίαση του καθηγητή Τίλεμανς είναι το θέμα των ε, δυνατοτήτων προτιμήσεων, δηλαδή να δοθεί επίσης προτεραιότητα στην οικογενειακή επανένωση και να ληφθούν υπόψη και διαφορετικές άλλες προτεραιότητες για να διευκολύνουμε την κοινωνική ενσωμάτωση. Και εδώ ερχόμαι στο θέμα της κατανομής των ποσοστώσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρξει ένα όριο για το κράτος μέλος. Πώς μπορεί να συνδυαστεί το συγκεκριμένο όριο και πόσο μπορεί να εντοπισθούν οι προτιμήσεις αυτές. Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα, το θέμα των πόρων για τη μετανάστευση με το οποίο ασχολείται και ο Ινιάτσιο Κοράος ασκιώδης εισηγητής. Δίνονται οικονομικές δυνατότητες στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει μια κάποια δυσκολία εδώ για να, να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι λόγοι ε, για τους οποίους δίδονται τα χρήματα αυτά και ποια είναι τα αποτελέσματα. Σαν παράδειγμα λέγεται ότι σε πολλές χώρες μέλη δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων και αυτών που αιτούνται άσυλο. Πρέπει να το δούμε αυτό, τα μέτρα αυτά πώς εφαρμόζονται και πόσο αποτελεσματικά είναι. Ευχαριστώ. Περνάω τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Παρακαλώ, 1,5 λεπτό το πολύ ο καθένας για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις και για να δευτερολογήσουν και οι συνεισηγήτριες. Παρακαλώ λοιπόν τηρήστε το χρόνο. Η κυρία Κιγιώμη είναι η πρώτη στον κατάλογό μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω γρήγορα δύο ομάδες ερωτήσεων για τους δύο ομιλητές μας. Πρώτη, σε ό,τι αφορά την πατέρα αρμοστή για τους πρόσφυγες, είπατε ότι το θεματολόγιο το ικανοποιεί και θέλει και τη βοήθειά μας. Είπατε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει ως το δυνατόν ε, περισσότερες νόμιμες οδούς. Η κλίδα κατανομής είναι το ερώτημά μου. Προτείνει η Κομισιόν για τη μετεγκατάσταση κάποιες κλίδες. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας. Σταθμίσεις κτλ. Δηλαδή πέραν των προτάσεων που έχουμε ήδη, αν ε, έχει νόημα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά ή όχι. Τώρα, ε, για τα private sponsorships σε κάποιες τρίτες χώρες όπως ο Καναδάς ή η Αυστραλία. Είναι μια νόμιμη ε, διάβλος, μια ασφαλή ε, δίωδος. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα για το αν και αυτό γίνεται σε κράτη-μέλη της Ένωσης ή όχι. Τώρα, στο δεύτερο μιλητή, τον κύριο Πόλετ, για το κοινό σύστημα ασύλου αν λειτουργεί αποτελεσματικά, έχουμε κάποιους ποιοτικού δείκτες για να βελτιωθούν τα πρότυπα υποδοχής και οι διαδικασίες. Η Κομισιόν εστίασε ε, στην πλήρη εφαρμογή των ε, προτύπων που μεταρρυθμίσαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μια αριστική προσέγγιση. Υπάρχουν όμως κάποια καινοτόμα μέτρα που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε για την εναρμόνιση των μέτρων. Και τέλος, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας με την αφορμή του κοινού συστήματος, ενημέρωση στη χώρα καταγωγής, ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτών κτλ. κτλ. Αν θέλουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εναρμόνιση, προς τα πού πρέπει να οδεύσουμε κατά την άποψή σας. Uh, now... Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σικόφσκι από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να σας ευχαριστήσω και για τον τρόπο που προεδρεύετε την ε, συνεδρίασή μας. Με πολύ ζωντανό τρόπο, πολύ ωραίο τρόπο. Το ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, τώρα, τους τελευταίους οκτώ μήνες. Το μόνο που κάνουμε, τουλάχιστον εγώ το μόνο που κάνω τους τελευταίους οκτώ μήνες, είναι να επισκέπτομαι κέντρα κράτησης, καταβλισμούς ε, ε, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες, ε, όπου ε, διαμένουν μετανάστες. Κάνω ό,τι μπορώ για να εξοικειωθώ με τα προβλήματα, με τα ζητήματα αυτά. Για να μην έχω αυτή την κοντόθωρη άποψη που μπορεί να έχει ένας κεντροευρωπαίος που φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Γιατί η Τσεχική Δημοκρατία δεν φαίνεται να αποτελεί χώρα στόχο και για πολύ χρόνο δεν θα γίνει χώρα στόχος ή χώρα προορισμού. Ιδίως λόγω των γλωσσικών φραγμών. Όμως, αν το δούμε σφαιρικά το ζήτημα, ε, σίγουρα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά τα ζητήματα. Και εμένα με απασχολεί το ζήτημα της ε, μετεγκατάστασης, μετακίνησης κτλ. Είναι λίγο, θα έλεγα, λαϊκίστικη αυτή η πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε 600.000 ε, ετούντες διεθνούς προστασίας ε, στην επικράτεια της Ένωσης για πέρυσι μόνο, το 2014. Και τα επόμενα δύο χρόνια Πόσοι θα μετεγκατασταθούν από αυτούς, μόνο 40.000. Κύριε καθηγητά, είναι αυτό ένα νούμερο αρκετό. Πείτε μας σας παρακαλώ, αν γίνει η μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων κάπου που δεν θέλουν να πάνε, θα μείνουν εκεί. Αυτό είναι ένα δικό μου προσωπικό ερώτημα. Εμείς, η οικογένειά μου κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από τα ε, σύνορα ε, έπρεπε να φύγουμε, έπρεπε να μετακινηθούμε. Φύγαμε, ξαναπήγαμε, ξανάρθαμε. Έχω εμπειρία λοιπόν από αυτή τη μετεγκατάσταση, προσωπική εμπειρία. Και δεν μας άρεσε και πάντα το μέρος στο οποίο πηγαίναμε. Πάντως χαίρομαι που θέσατε αυτό το ζήτημα για το κόστος. Ποιος θα επομιστεί το κόστος αυτό της μετεγκατάστασης. Έχω δει καταβλισμούς προσφύγων και έχω δει και τον τρόπο με τον οποίο φυλάσσονται και τον τρόπο με τον οποίο ε, πηγαίνουν τα, τα άτομα αυτά εκεί και πώς, σε τι συνθήκες διαμένουν. Τελευταία ερώτηση. Θέλουμε μια παγκόσμια, μια καθολική προσέγγιση και συστάση. Τι θα πει αυτό όμως. Ποσοστώσεις. Αυτό θα είναι η πανάκια κατά κάποιο τρόπο και θα χαλαρώσουν ως εκθαύματος όλες οι πιέσεις και το βάρος που αυτή τη στιγμή το απομίζονται Ιταλία και Ελλάδα κυρίως. Ευχαριστώ κύριος Ντούρεκ, είναι επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση ενέκρινε την εθελοντική υποδοχή μεταναστών. Η χώρα μου, η Πολωνία, πρόσφατα έχει απορροφήσει πολλούς πρόσφυγες και τις οικογένειές τους από την Συρία. Διάφορες οργανώσεις ασχολούνται με την επανεγκατάστασή τους. Έχουμε και την ευθύνη των περιφερειών σε διάφορες χώρες. Σήμερα μάλιστα μιλούμε για πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις χώρες του νότου της Ευρώπης και να έρθουν στην Ευρώπη και λόγω πολεμικών σειράξεων, αλλά όχι μόνο και διότι οι διακινητές γίνονται όλο και πιο δραστήριοι. Έχουμε λοιπόν απορροφήσει ήδη πρόσφυγες από την Τσετσενία, Τατάρους της Κρυμαίας και, δεν, και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτούς. Εμείς όμως τα κάνουμε αυτά στην ε, κεντρική Ευρώπη. Μην λησμονείτε ότι η κυριαρχία των κρατών είναι και κλειδί για τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να τα λησμονούμε αυτά. Καλά κάνουμε και τα συζητούμε αυτά τα πράγματα εδώ, αλλά όταν εξετάζουμε τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά δεν ανταποκρίνονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση προς τον κύριο Τέρκ του ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι ατυχές και μιλώ από τη σκοπιά της δικής μου χώρας για την ανθρωπιστική ε, στήριξη που προσφέρουμε επιτόπου στους ανθρώπους για να χρηματοδοτήσουμε και τη μαζική μετανάστευση προς την Σουηδία. Και μιλούμε για νόμιμη μετανάστευση. Υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Οι χώρες μέλη να υποδεχθούν κατά ποσοστώσεις τους μετανάστες. Έχουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Λιβύη που περιμένουν να περάσουν στην Ευρώπη. Ποιος θα επιλεγεί, αυτό θα γίνει σαλοταρία. Και εμείς οι Σουηδοί υποδεχόμαστε τους περισσότερους εδώ στην Ευρώπη. Και πρόκειται για τεραστίων διαστάσεων δυσκολία. Και γίνεται όλο και χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με την ενσωμάτωσή τους. Υφιστάμεθα βαρύτατες κριτικές στην Σουηδία. Τώρα για τον κύριο Τέλεμαν. Μιλάτε για 40.000. 40.000 μετανάστες τι γίνονται οι υπόλοιπε εκατοντάδες χιλιάδες που δεν λαμβάνουν άδειες παραμονής. Έχουμε αύξηση της τάξης του 100% των προσώπων που προσπαθούν να διέλθουν την Μεσόγειο. Τα σκεφτήκατε αυτά τα πρόσωπα. 40.000 ε, είναι ένα τίποτα. Ακούσαμε και για το σύστημα των ποσοστώσεων. και μας μιλάτε τώρα για επιβολή κυρώσεων για όσους ε, δεν δέχονται και ή δέχονται κτλ. Εμείς δεν αναγκάζουμε κανέναν, το κάνουμε από την καλή μας την καρδιά. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Κουά. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που παρακολούθησα σήμερα το πρωί, πολύ σύντομα τώρα, για την διαδικασία επαναγκαταστάσεως που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ το βρίσκω θαυμάσιο αυτό. Βεβαίω πρέπει να λάβει κανεί υπόψη, τα είπατε κι εσεί. Αυτή η ποσοτικοποίηση σε 20.000, αυτά πρέπει βεβαίω να, είναι, να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Τώρα για τι ποσοστώσει. Μου φαίνεται ότι αυτό που κάνατε ήταν πιο πολύ προβοκατόρικο όταν μιλήσατε για ανταλλαγή ποσοστώσεων ε, προσφύγων να μιλεί κανεί για ποσοστώσεις, ε, ποσοστώσεις πιο πολύ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν μπορεί να μιλεί κανεί για ποσοστώσεις για ανθρώπινα όντα και τα αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή η επανένωση οικογενειών, αυτά πρέπει να ληφθούν πολύ περισσότερο υπόψη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι το SR θα λαμβάνει υπόψη την εγκατάσταση σε κατά προτεραιότητα τοποθεσία. Σε ποια βάση όμω τώρα ο UNHCR θα κάνει τι αξιολογήσει αυτές. Επίσης έχω και μια παρατήρηση, άλλωστε τα είπαν και άλλοι πριν από μένα, για το γεγονό ότι πρέπει να εξετάσει κανείς όλες τις οδούς προσβάσεως τη μετανάστευσης και των προσφύγων και των ετούντων άσυλο που δεν υπάρχουν οι δύο διαυτές και πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανθρωπιστικές προξενικές θεωρήσεις. Βέβαια ο κ. δεν είναι εδώ αλλά να δούμε και τι κάνουν οι χώρες μας επιτόπου στις τρίτες χώρε, είτε στην Αίγυπτο είτε στην Τουρκία, για να διευκολύνουν τους πρόσφυγες. Ε, αρκούμε σε αυτά, αλλά βεβαίω όπω είπα πρέπει να γίνει μια συνολική προσέγγιση της ε, μετανάστευσης, όπως είπε και η κυρία Σίμπελ πριν από μένα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Λίγες ερωτήσεις τώρα. Πρώτο, πρόταση της Κομισιόν. Είναι αλήθεια ότι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, είναι βραχυπρόθεσμο μέτρο και αν εξετάσει κανείς καλύτερα το μέτρο, είναι περιορισμένο. Η στρατηγική δεν λαμβάνει υπόψη τις χώρες προέλευσης. Εκεί πρέπει να παίξουν ένα ρόλο και οι υπουργοί μας των εξωτερικών διότι εν τέλει πρόκειται για εξωτερική πολιτική. Περί αυτού μιλούμε εδώ. Θέλω να ακούσω τώρα και σχόλια από, για άλλα θέματα. Ο κύριος Τέρκ μίλησε πριν για μετανάστες που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και ιδίως για Σύρους και Ερυθρέους. Δεν λέει όμως τίποτα και τη διάκριση μεταξύ Ερυθρέων και Σομαλιανών. Τι γίνεται όμως και για τα πρόσωπα εκείνα που δεν προχωρούν από τη Συρία ούτε από την Ερυθρέα. Και όταν μιλούμε για επανεγκατάσταση, 20.000 άτομα σε δύο χρόνια. Αλλά μην λησμονούμε ότι μόλις τούτο το Σαββατοκύριακο πέρασαν την Μεσόγειο 5.000 άνθρωποι. Τι θα γίνει λοιπόν όταν θα εξαντληθεί το κατόφλι των 20.000, θα ξαναγυρίσουμε στο πρώτο τετραγωνάκι ο καθηγητής Τέλεμαν για τις κρίδες κατανομής και τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται, δεν θα πρέπει να περιλάβουμε και άλλα κριτήρια, για παράδειγμα το μέγεθος μιας χώρας, διότι αυτό το κριτήριο δεν έχει ληφθεί υπόψη για την εξέλιξη των κλειδών κατανομής. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Μάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Μου φαίνεται απλοϊκό να λέει κανεί ότι οι κλίδες κατανομής μπορούν να επιτύχουν την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Ένα που ζητεί άσυλο και τον στέλνουν στην Βουλγαρία, θέλει όμω να πάει στην Ολλανδία, στη Σουηδία, ε, δεν μπορεί, δεν θα το σταματήσει καμία κλίδα κατανομή. Και άλλωστε αυτό χαίρει και τη ελεύθερη διακίνηση μέσα στο, σύστημα Schengen. Για τον κύριο Τέλεμαν, πώ θα λειτουργήσει το θέμα αυτό. πώ θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Προεδρεύων κύριος Κίρκ Χοπ. Πρέπει να κλείσει ο κατάλογος ο κύριος Ντεπρέ. Εσείς ε, θα είστε όλη την ημέρα. Στην αρχή αναφέρθηκα στο θέμα σας για τις 4.30 το απόγευμα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνετε πάρα πολύ ώρα εδώ. Έχετε το λόγο. Είμαι προετοιμασμένος, Πρόεδρε γύρω από το σημερινό θέμα. Δύο σημεία. Είμαι υπέρ των νόμιμων τρόπων μετανάστευσης πρώτον. Είμαι υπέρ της ανθρωπιστικής θεώρησης και νομίζω ότι μια συνολική αντιμετώπιση της μετανάστευσης θα ενισχύσει τη θέση μας. Δεν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αγαθοί ε, δεν σημαίνει ότι αν ανοίξουμε νόμιμες πλευρές ε, θα καταργηθούν οι παράνομες και αν ε, δώσουμε θεωρήσεις ανθρωπιστικές αυτό δεν σημαίνει ότι θα καλύψουμε όλους έχουν ανάγκη. Δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί όπως είπα και το λέω αυτό σαν ανθρωπιστής. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τους ενδιαμέσους διότι οι ενδιάμεσοι επιταχύνουν τη ζήτηση και είναι και παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Δύο ερωτήσει στον κύριο Τίμερμαντς. Στο μηχανισμό κατανομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι μου κάνει εντύπωση. Η Ιταλία και η Ελλάδα θα επιλέξουν αυτούς οι οποίοι θα ανακατενεμηθούν επί τη βάση ποιων κριτηρίων. Ε, μήπως ε, τους πιο ενοχλητικούς θα τις στείλουμε στις χώρες υποδοχής και εμείς θα κρατήσουμε αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν τα λιγότερα από τα προβλήματα. Όταν σας άκουσα είχα και άλλη μια ανησυχία. Είπατε ότι τα κράτη τα οποία δεν θέλουν να υποδεχθούν αρκεί να πληρώσουν. Οπότε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ένα χρηματιστήριο ψυχών. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ πρέπει να υποδεχθώ 100 ε, αλλά δεν θα τους υποδεχθώ, θα πληρώσω μια άλλη χώρα να τους υποδεχθεί και έτσι θα αυξήσω την ε, προσφορά για τη χώρα αυτή, τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει περίεργες καταστάσεις μια τέτοια λογική. Τρίτον, για αυτούς οι οποίοι θα ωφεληθούν από την ε, μετεγκατάσταση. Τι είδου θεώρηση θα πάρουν, ποιο θα είναι το νομικό τους καθεστώς όταν μπουν στη διαδικασία της μετεγκατάστασης τι καθεστώς ε, θα απολάβουν. Εγώ είμαι υπέρ της ενίσχυσης Το budget de la Commission ΕΑΣΟ, ο προϋπολογισμός της ΕΑΣΟ δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ασθενής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σχεδόν οι οποίοι σεβάστηκαν το χρόνο που είχαν. Τώρα θα δώσουμε ίσα ίσα τον χρόνο στους ε, ομιλητές να δώσουν κάποιες απαντήσεις και μετά στους συνεισηγητές ε, ένα-δύο λεπτά ο καθένας. Πρώτον, η κυρία Κιέγκε... Ή μάλλον η συνεργάτης του κυρίου Τούρκ πρώτα θα δώσει ε, κάποιες απαντήσεις και μετά ο κύριος Τίμερμαντς. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Τρία λεπτά έχω για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Αδύνατο, ιδίω για έναν ακαδημαϊκό που έχει ώρες για, στη διάθεσή του. Θα ομαδοποιήσω τις απαντήσουν σε τρεις ε, κατηγορίες Ένα ερώτημα βασικό ήταν αν οι προτινόμενοι μηχανισμοί αρκούν πραγματικά, αν αποτελούν λύση ή ίσως και πανάκια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Φυσικά και όχι. Κανείς δεν το λέει αυτό άλλωστε. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σε σχέση με τα νούμερα, σε σχέση με την οικονομική αντιστάθμιση, την αποζημίωση που θα πάρουν τα κρατημέλη. Και άλλα μπορεί να σκεφτεί κανείς, άλλα κριτήρια, στάθμιση διαφορετική των κριτηρίων που συζητούνται επί του παρόντος κτλ. κτλ. Όλα αυτά νομίζω ότι ε, θεωρούνται δεδομένα και νομίζω όλοι συμφωνούμε από αυτού. Η προσωπική μου άποψη βέβαια είναι ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι να θεσπίζουμε μια σημαντική αρχή η οποία ζητεί περισσότερη πρακτική αλληλεγγύη και επιμερισμό ευθυνών. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να επιλύσουμε μια ανοιχτη τα προβλήματα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα σε σχέση με τη μορφή που έχει σήμερα. Και συμφωνούμε όλοι, νομίζω ότι δεν είναι καλό το σύστημα, όπως ισχύει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο σημείο ήταν οι δυνητικές καταχρήσεις του συστήματος. Δηλαδή, οι οικονομικοί μετανάστες ενδεχομένως ε, να είναι και δικαιούχοι αυτών των νέων μηχανισμών. Η πρόταση της Κομισιόν εδώ είναι σαφής. Λέει, οι οδοί αυτές, οι διάβλοι αυτοί ισχύουν μόνο σε αυτούς που έχουν ε, υπό περίπτωση πρίμα φάκες για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Πρέπει να έχουμε 75% ποσοστά αναγνώρισης ε, για τους επιλέξιμους ε, και ίσως και περισσότερο να είναι το ποσοστό. Άρα νομίζω ότι αυτό μπορεί κάπως να διασκεδάσει τις ανησυχίες ότι ίσως ανοίξει την πόρτα για καταχρήσεις αυτού του συστήματος και για μια αποτελεσματική εφαρμογή του σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή των ποσοστώσεων, ίσως και εμπορία ποσοστώσεων ως ακαδημαϊκός, εγώ ήρθα να σας αναφέρω τις διάφορες επιλογές που συζητούνται. Ποια είναι η προσωπική μου όμως άποψη. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ έχουμε αντιμετωπίσουμε πράγματι ε, ένα αντιστάθμισμα, μια, ένα δούνε και λαβή. Ξέρουμε ότι το Δουβλίνο δεν είναι αποτελεσματικό ο σύστημα από άκρος θεωρητική, αμυγός θεωρητική άποψη, αυτή η ανταλλαγή ποσοστώσεων θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν και μεγάλα μειονεκτήματα. Προσωπική μου άποψη λοιπόν, προς το παρόν, προς το παρόν ίσως οι συζητήσεις για εμπορία, για ανταλλαγή ποσοστώσεων μας αποπροσανατολίζουν από το τι θα ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε σήμερα. Εγώ δεν θα ήθελα ε, να αφήσουμε κατά μέρος ε, το θέμα του επιμερισμού ευθυνών. Δηλαδή κάποιοι να λένε ότι λόγω ανθρωπιστικών παραμέτρων δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό ίσως συζητηθεί στο μέλλον, δεν ξέρω. Πάντως, νομίζω ότι σε αδρές γραμμές οι προτάσεις της Κομισιόν είναι σωστές και πρέπει να θεωρηθούν ευπρόσδεκτες διότι, όπως είπα, εισάγουν μια σημαντική αρχή και αυτή μπορούμε να αναπτύξουμε στη συνέχεια περαιτέρω. Πρόεδρος. Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, ότι μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή ε, με ε, αν δεν έχουν απαντηθεί κάποια ερωτήματα. Το κύριος Πόλετ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δύο λεπτά πράγματι είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πάντως ευχαριστώ. Το θέμα της εφαρμογής τώρα και το πού βρισκόμαστε με τη μεταφορά στο διεθνές δίκαιο του πακέτου για το άσυλο. Δεν μπορώ να σας δώσω μια ξεκάθαρη εικόνα για τις 28 χώρες. Πάντως οι χώρες τις οποίες συμμετέχουν στην βάση δεδομένων Άιντα, η μεταφορά ε, είναι αργή σε πάρα πολλές χώρες. Η τελική προθεσμία είναι η 20 Ιουλίου 2015 και βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες είτε είναι στην φάση συζήτησης μιας πιθανής μεταρρύθμισης είτε συγγράφουν αυτή τη στιγμή ε, τις προτάσεις για την αλλαγή του συστήματος ασύλου του εθνικού. Πάντως αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά πολλούς τομείς, ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο. Απ' την άλλη έχετε χώρες οι οποίες είναι θα έλεγα πρωτοπόροι στη μεταφορά κάποιων από τις πιο περιοριστικές διατάξεις πριν γίνει δεκτό καν το πακέτο. Υπάρχει μια χώρα επίσης η οποία πριν τεθεί το θέμα της μετεγκατάστασης είχε ήδη εφαρμόσει και προσαρμόσει την ομοθεσία της σε σχέση με θέματα όπως η προσωρινή κράτηση. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το θέμα της μεταγκατάστασης και ποιους αφορά αν είναι αυτοί που είναι πρόσφυγες ή ήδη θεωρούνται πρόσφυγες ή αυτοί που έρχονται με θεώρηση ανθρωπιστικού τύπου. Αυτό εξαρτάται από τις εθνικές νομικές ρυθμίσεις, από το εθνικό δίκαιο. Και υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δίδουν ένα ειδικό καθεστώς ανθρωπιστικό, κάποιες άλλες επεξεργάζουν τους ανθρώπους αυτούς μέσα από τις εθνικές διαδικασίες και δίδουν επικορικού τύπου προστασία, αλλά οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές και αυτό υπογραμμίζει το ότι το παρόν καθεστώς προστασίας το οποίο χορηγείται επί τη βάση ακριβώς του κοινού συστήματος ασύλου ποικίλει, δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των θετικών αποφάσεων ε, για χορήγηση ασύλου. Κάποιες καινοτόμες προτάσεις για τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας έχουν γίνει, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το σύστημα δοκιμάζεται σαν παράδειγμα της κοινή επεξεργασίας αιτήσεων αυτό ανήκει έτσι και λιώς στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση που αφορά σε μια πρώτη κοινή επεξεργασία στηρίζοντας τις προτάσεις και των Ελλήνων και Ιταλών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα δουλέψει στην ουσία, πώς θα εφαρμοστεί πρακτικά. Ε, χρειάζεται αρκετή προσοχή βέβαια εδώ. Και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία έλεγα για τις διαφορές σε επίπεδο αναγνώρισης και για την ύπαρξη διαφορετικών ερμηνεών. Η Γαλλία σαν παράδειγμα έχει ένα ειδικό σύστημα αναγνώρισης για την Ερυθρέα 26% ενώ άλλες χώρες ξεπερνούν το 75%. ενώ όταν δούμε το ίδιο στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αν εφαρμοστούν οι ίδιες ποσοστώσεις, δεν ξέρω τι θα δώσει αυτό. Είναι θέματα, όπως είπα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν άμα τη εφαρμογή τους. Η εκπρόσωπος του κυρίου Τούρκ θα είμαι σύντομη γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο να επανέλθω σε κάποια από τα σημεία τα οποία τέθηκαν από αρκετούς από σας. Όπως είπε το κ. Στέρκ, αναφέρθηκε στην αρχική του δήλωση ότι υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετεγκαταστάσεις κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι αν εγκατασταθούν 40.000 άνθρωποι που θα έρθουν έτσι και αλλιώς στην Ευρώπη θα λύσουμε το πρόβλημα ή με το πρόβλημα με την εγκατάσταση 20.000. Δεν θα λυθεί το θέμα αυτών που έρχονται με παράτυπο τρόπο στην Ευρώπη. Και γι' αυτό απαιτείται το θέμα να αντιμετωπιστεί συνολικά. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται να δούμε βέβαια τις βασικές αιτίες που είναι στη ρίζα αυτού του φαινομένου και επίσης να δούμε τι γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσφυγες σε γειτονικέ χώρες για πολλά χρόνια όπως τη Συρία, την Κένια, την Αιθιοπία. Ε, να δούμε αν μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε και τις πρώτες χώρες υποδοχής είναι ένα πακέτο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι νομικές λύσεις είναι ένα τμήμα, πολύ σημαντικό, αλλά όχι το μόνο. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις για την ύπατη αυμοστία, για θέματα κοινή και ιδιωτικής κάλυψης δαπανών. Η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν ένα αναπτυγμένο σύστημα τέτοιου είδους και η Γερμανία στην περίπτωση των Σύρων έχει και αυτή κάτι το αντίστοιχο και αυτό ε, θα θέλαμε να το συζητήσουμε και να μοιραστούμε πληροφορίες για όσους από εσά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Για τα κριτήρια της μετεγκατάστασης, η ύπατη ασχολείται με το θέμα αυτό σε αρκετά κράτη-μέλη και σε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή όπως οι ανάγκες φυσικής προστασίας, εύθραυστες κατηγορίες, γυναίκες και άνθρωποι με ειδικά χαρακτηριστικά που χρήζουν περισσότερης προστασίας. Ε, επί τη βάση των κριτηρίων αυτών η ύπατη αρμοστία κάνει αν θέλετε τον πρώτο έλεγχο, αλλά οι τοπικές αρχές εμπλέκονται φυσικά και αυτές στη διαδικασία και δεν είναι αποκλειστικά η ύπατη αρμοστία η οποία επιλέγει αυτούς που θα προχωρήσουν σε μετεγκατάσταση. Να επανέλθω επίσης στις κλίδες κατανομής και τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εντοπίσει ορισμένα τέτοια κριτήρια. Μπορεί να γίνουν συζητήσεις και για τη συμπερίληψη και λήψη υπόψη και άλλων κριτηρίων για τις κλίδες κατανομής και το θέμα των προτιμήσεων των μεμονωμένων ανθρώπων αν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ή όχι. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο ως έχει. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις για το πώς και αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Αν το δει κανείς αυτό ε, για χώρες ε, κατάσταση όπως η Κένια, ε, τότε εκεί βέβαια οι προτιμήσεις ε, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχουν όμως ορισμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας όπως η οικογενειακή επανένωση και οι γλωσσικές, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά κτλ. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές πάντως έτσι ώστε να λάβουμε τις προτιμήσεις τους υπόψη. Αλλά αυτό λειτουργεί, οι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτή είναι μια ευκαιρία την οποία έχουν και ξέρουν τι τους περιμένει και πριν την εκκίνηση. Δεν καλύπτουμε πάντα τις επιθυμίες τους, αλλά εν πολλής νομίζω ότι το σύστημα είναι λειτουργικό. Σας ευχαριστώ όλους για να τελειώσουμε με αυτό το τμήμα της ημερήσιας διάταξης. Θα δώσω στις δύο συνεισηγήτριες να κάνουν μια μικρή παρατήρηση για να κλείσει η υπόθεση. Κυρία Μέτσολα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας σε συζητήσεις. Καλό θα ήταν να είχαμε και ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί στην ουσία συζητάμε τις προτάσεις τους. Πρέπει να τους προκαλέσουμε λοιπόν για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή σε μεγαλύτερο βάθος. Συμφωνούμε όλοι ότι πολλά πρέπει να γίνουν τελικά. αλλά τελικά σε πολιτικό επίπεδο οι πρωθυπουργοί θα πρέπει να συζητήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνώμη μας εδώ είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πολλά μένει να γίνουν να μας δοθούν κάποιες εξηγήσεις γιατί επελέγησαν δύο χώρες ε, υποδοχής, γιατί η Σομαλία δεν συμπεριλαμβάνεται, γιατί η Μάλτα δεν συμπεριλαμβάνεται. Επίσης, εγώ προέρχομαι από μια χώρα με υψηλό ποσοστό υποδοχής και χορήγησης ασύλου και θα δούμε ε, και με τη διαδικασία της μπλε κάρτας γιατί μόνο μία χώρα έχει ε, δεχθεί κάποιες ε, τέτοιου είδους ε, γιατί μια χώρα από 19.000 αιτήσει χορήγησε μία, ένα δικαίωμα ασύλου. Λοιπόν όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και να αναλύσουμε εκ νέου. Να συζητήσουμε επίσης και τα θέματα τα οποία έθεσε ο Φιλανδός συναδέλφος ε, γιατί σαν παράδειγμα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να επιλέξουν την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν και να μην υποχρεώνονται να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να τους λέμε ότι δεν θα μπορέσουν να τύχουν ασύλου. Εν πάση περιπτώσει οι χώρες οι οποίες δεν είναι στην περίγυρο της Μεσογείου δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι δεν έχουν ευθύνες. Ευχαριστώ κυρία Κέγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις ομιλίες τους, οι οποίες θα βοηθήσουν να βρούμε κάποιες λύσεις. Η προσπάθειά μας ε, περιλαμβάνει πάρα πολλές επιμέρους κατευθύνσεις, όπως είπε και η συνάδελφος, κυρία Μέτσολα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε περισσότερες εξηγήσει, περισσότερες λεπτομέρειες, για να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι θέματα τα οποία μένει να εμβαθυνθούν ακόμα, όπως η μπλε κάρτα, ε, θα ήθελα να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα κινητικότητας σε σχέση με την μπλε κάρτα, σαν παράδειγμα η κυκλική κινητικότητα που μπορεί να εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες. Είδαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μπλε κάρτα, αλλά δεν είναι το μοναδικό μέσο βέβαια για την αντιμετώπιση της οικονομικής μετανάστευσης. Ένα άλλο θέμα αφορά την αλληλεγγύη στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος για τον οποίο επελέγησαν δύο χώρες. Έχουν ε, δοθεί ε, κάποιες εξηγήσεις. Τώρα, γιατί όχι τους Ιρακινούς, γιατί όχι τους Λίβιους. Ε, όλα αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία τίθενται και θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς έτσι ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις. Κλείνοντας να πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και σε βραχυπρόθεσμες και σε μεσοπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες δράσεις. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε κάποιες διαρθρωτικές πολιτικές, να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τις ρίζες του φαινομένου και δεν αρκεί απλά να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ όλους για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους να σας πω πως ε, το επόμενο δίωρο ε, για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας είναι για τα τέλη Ιουνίου. Θα ορίσουμε ένα εισηγητή για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διαδικασία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Μέτσολα να δώσει τις εξηγήσεις που επιθυμεί. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει ελάχιστα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους ομιλητές και σας χαιρετώ και εγώ. mistake using her hammer. Uh, could you please... Uh, Ο πρόεδρος Κίρκ Χόπ. Σας καθ... καθίστε σας παρακαλώ γιατί ακόμα βλέπω πολλή κίνηση στην αίθουσα. Προτιμώ να κάθεστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Η κυρία Σαρτζεντίνη και άλλοι σας παρακαλώ. Μιας και απευθύνομαι προσωπικό σε εσά Καθίστε. Σας ανακαλώ στην τάξη κυρία Σαρτζεντίνη γιατί βλέπω ότι περιφέρεστε. Καλά λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση της τάξης των 5 λεπτών που δεν είναι και τρομερή βέβαια, αλλά να προχωρήσουμε για το επόμενο θέμα της ημερησία διατάξεως σήμερα είναι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για την καταπολέμηση απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με βάση το ποινικό δίκαιο. Δύο εισηγητές εν προκειμένου, Γκρέσλε, Ζίμπελ, ο τελευταίος τριμερής διάλογος για τη σχετική οδηγία έγινε στις 2 Ιουνίου. Συνεισηγητής είναι η κυρία Σίπελ που θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Οποιοςδήποτε ή οποιαδήποτε επιθυμεί να ε, κάνει ερωτήσεις κλπ. Μπορεί να το πράξει αμέσως μετά από την παρουσίαση της κυρίας Τζίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι βέβαια έξι τριμερείς διάλογοι βέβαια για μένα ήταν ο πρώτος. Ο έκτος λοιπόν τριμερείς διάλογος για την οδηγία PIF έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ε, βεβαίως με την διεύθυνση της κυρίας Γκρέσλε που είναι η συγκινητριά μας και με την εκπροσώπηση της μονίμου αντιπροσώπου της Λετωνίας τα πιο πολλά τεχνικά θέματα έχουν επιληθεί σε προηγούμενους τριμερείς διαλόγους. Άρα η συζήτηση στρέφεται τώρα γύρω από τα πιο ε, κέρια θέματα, δηλαδή απάτες σε δημόσιες προμήθειες, τα κατόφλια για ε, βαριά δικήματα και η συμπερίληψη του ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Όσον αφορά τούτο το, το λεγόμενο τελικό πακέτο, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος για τις ε, απάτες στις ε, δημόσιες προμήθειες και καταλήγουμε σιγά σιγά σε μια λύση. Για τα άλλα θέματα ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τις κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων το Κοινοβούλιο θέλει τουλάχιστον ανώτατη ε, ποινή, ε, μάλλον κατώτατη ποινή 5 ετών και 15.000 ε, ευρώ κύρωση χρηματική. Τέσσερα χρόνια για το Συμβούλιο και 100.000 μη δεσμευτική βέβαια χρηματική ποινή. Εμείς μπορούμε να δεχθούμε τέσσερα χρόνια ποινή και να αυξηθεί το όριο της χρηματικής ποινής στα 100.000 ευρώ, αλλά θέλουμε το όριο ποινής να είναι δεσμευτικό. Το Συμβούλιο δεν το δέχεται αυτό για την περίοδο παραγραφής, για την δίωξη. Εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε μια ενιαία περίοδο παραγραφής της τάξης των 5 ετών. Το Συμβούλιο δεν δέχεται τον κανόνα αυτό χωρίς εξαίρεση για τις χώρες εκείνες μέλη όπου οι εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν αναστολή της διώξεως. Εν προκειμένου, Υπάρχει βέβαια μια βάση για συμβιβασμό, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την τελική δέσμη μέτρων. Ε, επιβολή κυρώσεων το Κοινοβούλιο ζητεί περίοδο 10 ετών, το Συμβούλιο 5 ετών. Τώρα, συμβιβασμό σε 7 ή 8 χρόνια προτάθηκε μεν από το Κοινοβούλιο, δεν έγινε όμως δεκτό από το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν τώρα, εκτός από αυτό, μένει και ο ΦΠΑ που είναι το πιο επίμαχο θέμα. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να περιληφθεί ο, ο ΦΠΑ μέσα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Το Συμβούλιο όμω είναι απολύτω αντίθετο με τη συμπερίληψη του ΦΠΑ και δεν προβλέπεται τουλάχιστον για την ώρα καμιά συμβαστική λύση. Ήταν λοιπόν ο τελευταίος τριμερής διάλογος υπό ε, Λετωνική Προεδρία και τώρα βέβαια αναμένουμε την επικείμενη Λουξεμβουργική Προεδρία όπου ελπίζουμε ότι θα μπει κάποια φρέσκια ε, ενεργητικότητα και βεβαίως, βεβαίως ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ που ε, για μας είναι ασφαλώς το πιο σημαντικό πράγμα για το κοινοβούλιο, το πιο σημαντικό θέμα για το κοινοβούλιο. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος Κίρκ Χοπ. Ευχαριστώ. Ε, σε βάθος ανάλυση και πάρα πολύ χρήσιμη. Βλέπω ορισμένου σκιώδη συγητά ή συγητρία. Δεν είστε υποχρεωμένε να μιλήσετε, αν θέλετε. Νομίζω ότι οι εξηγήσει και Ζήπερ υπήρξαν πολύ πλήρε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τότε α προχωρήσουμε και έχουμε και μάλιστα ένα κέρδο δύο λεπτών ή τριών. Δεν θα διακόψω βέβαια για τα δύο λεπτά. Μπορούμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στο επόμενο θέμα. Α, με συγχωρείτε, ναι, διακόπτε Εγώ θα το πράξω όμω και σωστά, σύμφωνα με τι σημειώσει που έχω μπροστά μου. Θα πρέπει να πω λοιπόν αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Κίρκοπ, που είναι εισηγητής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ έχει συντάξει νέα ε, εκδοχή του, της, ε, του σχεδίου ένα σημαντικός αριθμός 787 τροπολογιών και που αναφέρονται σε όλα τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, δηλαδή άρα όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ίδια την έκθεση και θα διεξαχθεί ανταλλαγή απόψεων. Έχουν γίνει τρεις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Εγώ πρώτα ως πρόεδρος θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Κίρκχοπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, απευθύνω στον εαυτό του κύριο Κίρκχοπ. Ως πρόεδρος, ε, όπως μάλιστα όπως είπατε ως πρόεδρος, ε, υπάρχει ένας αριθμός τροπολογιών ε, που έχουν υποβληθεί για την έκθεσή μου. Ο αριθμός τους, ο υψηλός αριθμός τους δείχνει και πόσο σημασία αποδίδουν στην έκθεσή μου οι συναδελφοί μου. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέχρι τέλους του έτους ή δυνατόν. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι άλλοι θα τονίσουν ότι υπάρχει επιθυμία να διεξαχθεί πρόοδος για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων ταυτόχρονα. Υπάρχει λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή κάποια κίνηση και αυτό με ενθαρρύνει. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε την θέση μου έως τώρα, ότι πιστεύω δηλαδή ότι η οδηγία δεν είναι μονάχα ουσιώδης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και εγκληματικότητας, αλλά διότι πρέπει να περιλάβει και τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία δεδομένων και την επεξεργασία τους, καθώς επίσης και αποζημίωση ε, προσώπων ή ατόμων για ιδίως επιβάτες. Θέλουμε να προστατεύσουμε ζωές, θέλουμε να προστατεύσουμε και τις ε, δημόσιες ελευθερίες και αυτά μπορούν να συμβαστούν μέσα στην οδηγία. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουμε λάβει, αυτές καλύπτουν ευρύτατο φάσμα. Ε, οι διάφοροι ευρωβουλευτές ξεκινούν από το να ζητούν την απόλυτη απόρριψη της οδηγίας και βεβαίω και αναφέρονται και στην ε, κοινοποίηση ε, δεδομένων μεταξύ χωρών και ούτω καθεσής. Εγώ έχω καταστήσει σαφή την ε, θέση μου στην αναθεωρημένη μου έκθεση, αναθεωρημένη επισημένο έκθεση, διότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρονται ακόμα μονάχα στις προτάσεις της Κομισιόν και αυτό από την κοινοβουλευτική άποψη είναι απολύτως απαράδεκτο. Έχω απόψεις και βεβαίως για κάθε μια από τις τροπολογίες, αλλά προτιμώ να εξηγήσουν τις απόψεις τους ή καταθέτονται στις τροπολογίες, διότι βεβαίω είμαι και παγιδευμένος εδώ στον προεδρικό φόκο σήμερα, υπάρχουν πάντως κάποια βασικά στοιχεία όπου μπορούμε να επιτύχουμε συμβιβασμούς. Αυτά τα βασικά στοιχεία είναι οι διατάξει για την προστασία των δεδομένων και σχετικές ρήτρε προφύλαξη και καλύτερη κοινοποίηση των δεδομένων, καθώς και κανόνες που να διέπουν την κοινοποίηση αυτή μεταξύ χωρών, διαβίβαση μεταξύ χωρών των δεδομένων. Και επίσης όταν ε, επιβάλλουμε μέτρα, νομοθετικά μέτρα για την χρήση των προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζεται ότι θα γίνεται και αυτή η κοινοποίηση στη βάση της αποτελεσματικότητας και τα εργαλεία που προτείνουμε να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται ορθά. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν νομοθετικέ δυνατότητε, τι οποίε δεν χρησιμοποιούν ή πάντω δεν χρησιμοποιούν σωστά οι χωρισμένοι. Αυτό το θέμα όπω είπα περιλαμβάνεται βεβαίω και σε πολλέ από τι τροπολογίε. Νομίζω ότι έχουμε συλλέξει σημαντική εμπειρία εδώ σχετικά με σημαντικά μέτρα τα οποία περνούν και τα οποία έχουν ενισχύσει την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου. Ορισμένοι εξημών βεβαίως έχουμε απογοητευτεί τα τελευταία χρόνια διότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως θα έπρεπε και με τον κατάλληλο, με τον ορθό τρόπο. Μπορούν να περιληφθούν και άλλα δικήματα στο πεδίο εφαρμογή της οδηγία καθώς και η συλλογή δεδομένων όχι μόνο για πτήσει εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για πτήσει εντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ξεκάθαρη. Εφόσον υπάρχουν οι μηχανισμοί αναθεώρησης των ε, οδηγιών αυτών θα πρέπει να φτιάξουμε μια νομοθεσία που να μην επιτρέπει παραθυράκια που να μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίε. Οι ισχυρότεροι ηγητέ και εγώ προσωπικά έχουμε συναντηθεί κατά επανάληψη και νομίζω προσπαθήσαμε όλοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Ωστόσο είμαι ρεαλιστή και αισιόδοξο άνθρωπο. Και ελπίζω ότι θα επιβιώσω και τη σημερινή συνεδρίαση. Συμφωνούμε σε όλα μέχρι τώρα. Όχι. προφανώ όχι. Θεωρούμε ότι θα είναι εύκολη υπόθεση η οδηγία αυτή. Πάλι όχι. Πιστεύω όμω ότι προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κοινέ λύσει με στενή συνεργασία. Και ελπίζω ότι σύντομα θα επανέλθουμε στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα όπου θα μπορούν να το υποστηρίξουν η πλειοψηφία των πολιτικών μα ομάδων και μελών μα. Είμαι βέβαιο ότι χρειάζεται αναλογικότητα του συστήματο και είμαι βέβαιο επίση ότι απαιτείται μια λύση ταχεία το, στο αυτό συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, οι χώρες μέλη, οι αρχές επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικές και απαιτείται να εξεύρουμε τις ορθές λύσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους εκείνους που μας παρέσχουν πληροφορίες και κατευθύνσεις που απάντησαν πολλές ερωτήσεις, καθώς επίσης ευχαριστώ για το ότι έθεσαν υπόψη μας τη σχετική τους τεχνογνωσία. Ευχαριστώ και τους και ηγητάς και εισηγητρίας που έχουν δουλέψει πραγματικά σκληρά και έχουν συνεργαστεί πλήρως και μαζί μου για να προωθήσουμε την οδηγία, την έκθεση δηλαδή. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους μου για να μπορέσουν να αναπτύξουν τα επιχειρηματά τους. Ο Άξελ Βος δεν είναι παρόν σήμερα, αλλά εκπροσωπείται με θαυμάσιο τρόπο από τον κύριο Ντία Στεμέρα που θα μιλήσει και πρώτος εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, μιλάω εξ ονόματο του Άξελ, ο σκιώδη ε, της τη σημαντική αυτή έκθεση. Και θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω ω συζητητή για την εντατική και αποτελεσματική δουλειά που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Ο Άξελ είναι στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ήθελα να σας μεταφέρω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια στη Ρήγα εξέφρασαν τεράστια ανησυχία για την βραδύτητα που επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ομοθετικής πρότασης για το PNR, το Ευρωπαϊκό PNR. Τώρα θα ήθελα να, εφαρμοστώ, να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Το ΕΛΚ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το συντομότερο δυνατό να τοποθετηθούμε με στόχο να ξεκινήσουν οι διοργανικές συζητήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Το Κοινοβούλιο νομίζω ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά. Έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που κατατέθηκαν τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κύρκο. Ο εισηγητής κάνει εξαιρετική δουλειά, το προείπα και το παραλαμβάνω. Ωστόσο, Έχουμε συνεδριάσει μέχρι και πέντε φορές οι σκιώδεις, δυστυχώς όμως χωρίς να σημειώσουμε καμία πρόοδο. Συζητήσαμε τα άρθρα 7, 7α, 8 και 1, όμως επιμένω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα. Θέλω να επαναλάβω ποια είναι τα σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόκειται για σημεία των οποίων ε, δεν είμαστε διτεθειμένοι να κάνουμε πίσω. Γιατί, γιατί για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των πολιτών μας από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλα σοβαρά εγκλήματα ή σοβαρές αξιόπινες πράξεις. Ε, έχουμε καταθέσει 70 τροπολογίες ε, ως Έλκ για τα βασικά αυτά σημεία. Τι ζητούμε λοιπόν ουσιαστικά, το λέω για να είναι σαφές. Πρώτον, επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Εμείς θέλουμε να συμπεριληφθούν οι ενδοκινοτικές πτήσεις και οι εθνικέ πτήσεις, εσωτερικού να συμπεριληφθούν επίσης ώστε παραβάτες ή ε, ε, ξένοι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτά. Δεύτερον, να, να έχουμε και τους ε, τουριστικούς φορείς που πουλάνε ταξιδιωτικά πακέτα και πτήσεις τσάρτερ τα στοιχεία PNR των πελατών τους τα ε, συγκρατούν μένα, αλλά δεν τα δίνουν απαραίτητα στην αεροπορική εταιρεία. Πρέπει όμως να δίνονται αυτά τα στοιχεία PNR σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πρέπει να σας πω ότι η ίδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου απεφάνθη και μάλιστα θετικά. Τρίτον, ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Europol Τη Ευρωπαϊκή αστυνομία. Δεν ε, επεκτείνουμε, αλλά είναι κάτι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό. Ζητούμε ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ. Δεν θέλω να επεκταθώ όμω. Περίοδος διατήρησης και κρυπτογραφημένα στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικό για την περίοδο διατήρησης των στοιχείων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν διατηρούνται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτά τα στοιχεία και ξέρω γιατί μιλάω, σας το λέω, αυτό σημαίνει ότι οι έρευνες δεν θα φέρουν, δεν θα δώσουν καρπούς. Ιδίως όταν υπάρχουν κυκλώματα που σταματούν ακριβώς προσωρινά τις δραστηριότητες τους σκοπίμως για να χαθούν τα ίχνη τους. Και μετά ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι με μεγαλύτερη ομότητα και βία πιο μετά. Το ΕΛΚ ζητά επιμήκυνση ε, του χρόνου διατήρηση των στοιχείων από τα 4 στα 7 έτη. Μετά την 7η ετία θα πρέπει μονίμως να διαγράφονται, να καταστρέφονται αυτά τα στοιχεία. Ε, κρυπτογράφονται μετά από έξι μήνες ε, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευαίσθητα στοιχεία. Ναι, για να είμαστε αποτελεσματικοί και να έχουμε μια ψηλή προστασία για τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική αρχή εποπτείας. Θα είναι ανεξάρτητη αυτή η αρχή σε κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει να υπάρχει και ένας αρμόδιος προστασίας ε, για τα στοιχεία PNR που ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, αξιολογεί και να συντονίζει την επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Τώρα, κατάλογος σοβαρών αξιόπινων, σοβαρών αδικημάτων Ποια είναι αυτά τα σοβαρά ε, αδικήματα. Θέλουμε, και το έχουμε στην τροπολογία 277, ε, θέλουμε να υπάρχει ένα κατάλογος, μία λίστα για όλα τα αδικήματα, όλες τι αξιόπινες ε, πράξεις που αποτελούν απειλή για τη δημόσια γνώμη. Υπάρχει ένα γαλλικό παράδειγμα. 3 Ιουνίου, ο Ντόι Σετσάιτον μα είπε ότι ε, και η δεξιά και η αριστερά στη Γαλλία ζητά ε, ταχεία πρόσβαση στα στοιχεία και δει τα στοιχεία PNR για αυτούς που ερευνούν περιπτώσεις τρομοκρατίας. Και στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση μια εξεταστική επιτροπή αναφέρθηκε στην περίπτωση της απώλειας των λιχνών του Σαντίχ Κουασί που είναι ένας, ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης, του Σαρλί Εμπτό, όταν είχε πάει από τη Παρίσι στη Γάνς αν αργεί πάρα πολύ, ε, η, αν αργεί ακόμη περισσότερο η συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό PNR, ή αν είναι πολύ περιοριστικό, οι Γάλλοι από μόνοι τους ε, θα συνάψουν ε, συμφωνίες διμέρης για την ανταλλαγή στοιχείων PNR. Και κατά πάσα πιθανότητα λένε Ε, θα είναι πολύ, λιγότερο, πολύ λιγότερες οι ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με το ευρωπαϊκό πιάνο και ίσως το κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό μεμονωμένα εάν δεν μπορέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εγκριθεί αυτό το ε, ευρωπαϊκό PNR. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ακούσουμε, να εισακούσουμε τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε συμβιβαστικές προτάσεις. Αυτή είναι η άποψη του ΕΛ και αυτή είναι η άποψη και η δική μου αλλά και η άποψη του Άξελ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από αυτή την πραγματικά θαυμάσια εξέταση του θέματος. Πού να αρχίσω άραγε. Βέβαια όλοι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν ξέρω τώρα αν πρόκειται για μεταφραστικό αμάρτημα, αλλά άκουσα στην μετάφραση να μου λένε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απαιτεί. Βεβαίως όλοι μπορούμε να απαιτούμε, αλλά εν τέλει όλοι καλούμεθα να συμβιβαστούμε και αυτό νομίζω ότι αποτελεί και την βάση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Παρόλες τις διαφορές και με παραπάνω από 700 τροπολογίες. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να βάλει την βάση για μια κοινή συζήτηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ξεκάθαρους συμβιβασμούς. Συζητούμε με τον ε, πρώτο εισηγητή βεβαίως ήταν σύντομες οι συναντήσεις διότι δεν διαθέταμε τις μεταφράσεις των τροπολογιών και δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε επομένως τις επιμέρους τροπολογίες. Άλλωστε, γρήγορα δεν σημαίνει και καλά. Θέλω να επισημάνω και πάλι το ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε από κοινού ως Κοινοβούλιο και όπου συμφωνήσαμε ότι θέλουμε ή δυνατόν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό PNR σύστημα δηλαδή καταγραφή των προσωπικών δεδομένων των επιβατών ε, αεροπλάνων. Το θέλουμε να μπει ως τμήμα του πακέτου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν μιλεί το Λαϊκό Κόμμα για προστασία των πολιτών, βεβαίω, είναι σημαντικό να προστατευτούν οι πολίτες από αδικήματα, από ποινικά αδικήματα. Ορισμένοι όμω, ε, μάλλον 99,9% λένε ορισμένοι, 99,9% των πολιτών των οποίων συλλέγονται τα ε, δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα όταν μεταβαίνουν κάπου με αεροπλάνο, είναι αθώοι πολίτες. Επομένως δεν πρέπει να καταλήξουν, να πέσουν μέσα στα γρανάζια κάποιων συστημάτων, ορισμένοι από τους πολίτες αυτούς, λόγω ενδεχόμενης εσφαλμένης χρήσης των δεδομένων τους. Αυτό ισχύει βεβαίως και για τον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων. Εγώ οτιδήποτε αποτελεί απειλή πρέπει να μπει στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων, λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν εκεί οι απειλές και όπου τα PNR προσφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία. Μπορούν να υπάρχουν και αδικήματα όπου η συλλογή των PNR να μην προσφέρει απολύτως καμιά προστιθέμενη αξία. Εκεί τότε παραπλανούμε τους πολίτες λέγοντας ότι ε, σε κάτι συμβάλλει η συλλογή των PNR. Εκεί χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικέ. Πρέπει βέβαια να σκεφτούμε, και το είπαμε αυτό και στο ψήφισμα, με ποιον τρόπο δηλαδή μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο το, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και να δημιουργήσουμε και την ασφάλεια ότι δεν θα επαναληφθούν πράγματα όπως με την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και όπου νομίζω ότι υπάρχει ο σχετικός φόβος. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε και το πιο σωστό είναι να καταβάλουμε προσπάθεια για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής αλλά και τις περιόδους αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων Εφόσον οι εγκληματίες αναμένουν να παρέλθουν οι προθεσμίες διατηρήσεως των δεδομένων πριν να προβούν σε νέα αδική πράξη, σε νέα ποινικά αδική πράξη δηλαδή, ε, τότε ας το βάλουμε την περίοδο, το λέω ειρωνικά βέβαια αυτό, σε μια τάξη 50 ετών, ώστε να μην ξανακάνουν ποτέ τίποτα. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα επιβατών διαμεθοριακών πτήσεων. Εάν κάποια στιγμή μας ξεφύγει τέλο πάντων ένας εγκληματίας, ένας εγκληματίας που έχουμε ή τα χαρακτηριστικά της εμφάνισής του ή και το όνομά του, θα δούμε ποια είναι η πραγματική αξία του PNR. Εάν έχω τον, το όνομα ενός εγκληματία, τότε βεβαίως υποθέτω ότι έχουμε πλήθος μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως και το σύστημα API, για να βρούμε τον δράστη αυτόν. Η ιδιαίτερη αξία των δεδομένων PNR είναι έγκυται στο ότι με τη σωστή χρήση αλγορίθμων μπορούμε να αποκαλύψουμε δράστες ποινικών αδικημάτων των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη βεβαίως και στη συζήτηση των τροπολογιών. Εν τέλει έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις σε πολλούς τομείς Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι μπορούμε ε, να ε, πορευτούμε σε έναν καλό δρόμο, σε μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά σημεία. Για μας, ξαναλέω, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υψηλό επίπεδο προστασίας, υποχρεωτική χρήση των ε, συστημάτων και βεβαίως να διασφαλίσουμε ότι εν τέλει, αυτό αποτελεί άλλωστε και την επιθυμία του Συμβουλίου που μας υπέβαλε, εν λοιπόν, να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη και όχι 28 ή και 29 πολύ διαφορετικά συστήματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και είμαι πεπισμένη έστω και αν δεν μπορώ να σας δηλώσω τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σοφίντφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και εισηγητά, ταυτοπροσωπεία. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την Birgit, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό έχει μια ιστορία ταραγμένη μέχρι τώρα. Και είναι καλό που έχουν ξαναρχίσει οι διαπραγματεύσεις σε επικοδομητικό πνεύμα. Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Διάς γιατί αυτά που είπε δεν αντικατοπτρίζουν τις διαπραγματεύσεις τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι η παρατήρηση ότι το Κοινοβούλιο κολυσιεργεί στο θέμα PNR δεν έχει καμία δικαιολογία. Θα ήθελα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου να μας πούν πότε αυτοί σκοπεύουν να κάνουν τις τελικές τους προτάσεις. Αυτή τη δεκαετία, καλό θα ήταν να το ξέραμε. Εγώ περιμένω εδώ και δυόμισι μήνες για μία απάντηση σε μία επιστολή. Και δεν ξέρω αν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου στείλει με περιστέρι ταχυδρομικό την απάντηση αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Το θέμα της επιστολής μου είχε δύο θέματα βασικά. Καταρχάς, πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, τις οποίες δεν πήρα καμία απάντηση, σχετικές με την ανάγκη της αναλογικότητας του ε, προγράμματος Ευρωπαϊκού PNR. Και δεύτερος, με την πολύ καθυστερημένη πλέον νομική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της απόφασης για την παρακράτηση των στοιχείων, των προσωπικών στοιχείων. Κανονικά πρέπει το θέμα αυτό να κλείσει πριν το τέλος του χρόνου. Ε, περιμένω όμως την Επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί αν δεν κάνουν κάτι αυτοί δεν θα κάνουμε κι εμείς. Χρειάζεται να παίζουν όλοι το παιχνίδι για να προχωρήσει. Ελπίζω να με καταλάβατε. Μία επιπλέον παρατήρηση πριν μπω στα θέματα ουσίας. Η πρόταση του κυρίου Διαστεμέρα από πλευράς του ΕΛΚ ότι θα είχαμε αποφύγει το Σαρλί Εμπτό αν υπήρχε το PNR. Αυτό είναι σαν χλαμάρες κύριε Έδιες και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω. Αλλά το να αρχίσουμε τώρα να λέμε αν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό PNR αν είχαμε δηλαδή καταπιεί την πρόταση την προηγούμενη χωρίς συζήτηση δεν θα υπήρχε επίθεση στο Σαβλί Εμπτό. Αυτό είναι πραγματικά αποκρουστικό σαν πρόταση. Λοιπόν, για τη δική μου πολιτική ομάδα υπάρχει μία βασική προτεραιότητα. Το πώς εμείς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ε, τον διαμοιρασμό των πληροφοριών. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για την παρακράτηση των προσωπικών στοιχείων, αλλά μιλάμε για τη χρήση των στοιχείων αυτών για πρακτικούς λόγους από διαφορετικούς φορείς. Αν τώρα τα δεδομένα αυτά γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από 28 διαφορετικούς οργανισμούς, δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει υποχρεωτική και ε, κατανομή των στοιχείων, να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων PNR, αλλά να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για, τον τρόπο, για τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε μια συνεκτική πρόταση. Εμείς είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος και μίας ενιαίας μονάδας ευρωπαϊκής επεξεργασίας και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως μέσω κανονισμού και όχι τόσο μέσω οδηγίας. Αλλά τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις συζητήσουμε αν και το σημείο αυτό είναι κομβικό. Τώρα, για την εμβέλεια, τις ρήτρες ασφαλείας και τα λοιπά, όλα θα εξαρτηθούν από το ποιο θα είναι το πρότυπο της μονάδας αυτής, το πρότυπο λειτουργίας εννοώ της μονάδα αυτής για την εμβέλεια. Μιλάμε τώρα για ένα κατάλογο ποινικών πράξεων που θα πρέπει να καλύπτονται. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, αλλά καλό θα είναι να συμπεριλάβουμε επίσης και την δυνατότητα αναθεώρησης αυτού του καταλόγου, γιατί ο κόσμος αλλάζει, υπάρχει μια δυναμική διεθνής. Δεν έχουμε συγκεκριμένες εμπειρίες με ένα τέτοιο σύστημα, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε αν το PNR πράγματι συνεισφέρει στην πρόληψη ή την επίλυση τέτοιου είδους ποινικών πράξεων. Και κάποιες από αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν, κάποιες θα πρέπει να προσθεθούν. Οι ρήτρε προστασία δεν θέλω να περάσω στην παρούσα φάση σε λεπτομέρειε, αλλά καλό θα είναι το Συμβούλιο να μα δώσει στοιχεία για την οδηγία προστασία των προσωπικών δεδομένων για τις ενδοκινοτικές πτήσεις ή τις άλλες μορφές μετακίνησης θα διαφωνήσω. Ε, εμείς είμαστε κατά τη συμπεριλήψη των ενδοκινοτικών μετακινήσεων ή άλλων μορφών μεταφοράς. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμα από την Birgit Σίπελ, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε, είναι η στόχευση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού, ε, να περιορίσουμε δηλαδή όσο μπορούμε περισσότερο τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων και τη χρονική διάρκεια της περίοδου παρακράτησης. όχι πάνω από 30 ημέρες, μετά από τις 30 μέρες θα διαγράφονται, εκτός αν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα βέβαια θεωρούνται και κρίνονται απαραίτητα για μια συγκεκριμένη έρευνα. Αλλά για να μπορέσουμε πράγματι να πάρουμε αποφάσεις πάνω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, απαιτούνται οι πληροφορίες που έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χιλιάδες φορές και δεν μας έχει δώσει. Δύο τελικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Διαστεμέρα. Είπατε ότι θα πρέπει να ακούμε το τι λένε τα εθνικά κοινοβούλια. Κοιτάξτε, πρώτα θα πρέπει να πάρουμε μια θέση και μετά αφού έχουμε τη θέση θα διαπραγματευτούμε. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το αντίθετο. Πρώτον λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε και στη συνέχεια, και δεν είναι τόσο εύκολο όπως είπε και ο εισηγητής, Νομίζω ότι είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι στόχοι κοινοί. Δεν λέγω ότι υπάρχει εγγυημένο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2015, αλλά είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η επιτυχία μας όμως θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια την οποία θα κάνουν όλες οι πολιτικές ομάδες και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ Σοφή Άλμπρεχτ. Thank you Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλές από τις κριτικές παρατηρήσεις. Να απαντήσω πρώτα στις απαντήσεις του Δίας Τεμέρα. Η έκφραση που χρησιμοποίησε ότι παράληψη συλλογής δεδομένων οδηγεί σε βία και έγκλημα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πώς θα αποτρέψουμε κάποιους από το να κάνουν βίες κλιματικές ενέργειες με τη συλλογή δεδομένων. Αυτά γίνονται με πρόληψη, με τη δημιουργία μιας κοινωνίας που να οδηγεί σε χαμήλωμα των επιπέδων της εγκληματικότητας. Αυτά λέει η εγκληματολογία. Δεν λέει για ε, συλλογή δεδομένων. Αν θέλουμε δηλαδή να βρούμε λύσεις πραγματικά για ασφάλεια και για να ρίξουμε τα επίπεδα της εγκληματικότητας που αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος τελικά. Δεύτερο, οι εγκληματίες πάνε και βρίσκουν τα παραθυράκια. Αυτό ακούω. Βεβαίως, εδώ συμφωνώ με την Μπίρκετ Ζίπελ. Τι σημαίνει αυτό, χρειαζόμαστε πλήρη κάλυψη τότε γιατί δεν κρατάμε και για 100 χρόνια τα δεδομένα, διότι μπορεί αυτοί να επανέλθουν πολλά χρόνια αργότερα. Να γνωρίζουμε τι έχουν κάνει και πριν από 20 χρόνια για να έχουμε πλήρη κάλυψη. Επίσης, γιατί δεν κρατούμε τότε και τα δεδομένα των επιβατών του σιδηροδρόμου. Εγώ μπορώ να πάρω την, ε, τους γερμανικούς σιδηροδρόμους και να ταξιδέψω σε όλη την Ευρώπη ανώνυμα. Μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο. Γιατί τότε δεν ελέγχουμε και τον τελευταίο επιβάτη αυτοκινήτου. θέλετε πλήρη κάλυψη, τότε αυτά πρέπει να κάνετε. Και βέβαια οι δημόσιες μεταφορές, ακόμα και τα ποδήλατα. Θα έχουμε και διασυνδεμένα ποδήλατα σύντομα. Connected bikes Αυτά θα πρέπει να περιλάβετε τότε στα, στην ατζέντα σας. Και αυτά είναι που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που το έκρινε παράνομο με την απόφασή του για την Data Retention Directive πέρσι τον Απρίλιο. Πάνω από ένα χρόνο λοιπόν είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου και σε μια κοινωνία όπου έχουμε και των χάρτη μερικών δικαιωμάτων, προστασία της προσωπικής σφαίρας κτλ. Κάθε φορά που αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα εννοώ βέβαια έτσι, χρειαζόμαστε τουλάχιστον κάποια αναλογική διασύνδεση με τουλάχιστον μια υποψία. Δεν μπορείτε να βγείτε και να συλλέγετε τα δεδομένα όλων επειδή δεν ξέρετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Πρέπει να βρείτε καλύτερες λύσεις. Χρειάζεται απειλή χρειάζεται υποψία. Αυτό είναι κλασική αστυνομική δράση. Εκεί έχουμε και την ε, πρώτη ε, τροπο, τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν μπορείτε λοιπόν να χωθείτε παντού. Τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό πρέπει να τηρήσουμε. Και για τούτην εδώ την αδικία η οποία προτάθηκε μάλιστα πριν από την έκδοση της ε, αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αυτή λοιπόν η οδηγία δεν προβλέπει καμιά δικαιολόγηση σχετικά με το ποιε πτήσεις είναι ενδεχομένως ε, έχουν, περιέχουν κάποιο ρίσκο, ούτε σε ποιες περιοχές, ούτε για τους επιβάτες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία και για την ε, καταγραφή του προφίλ του κάθε επιβάτη. Γίνεται αυτόματα και για πάντα. Δηλαδή συλλέγουν στοιχεία του προφίλ του κάθε επιβάτη και για πάντα. Μα αυτό δεν σημαίνει στόχευση. Δεν υπάρχει ούτε καμία ανάγκη έγκρισης τουλάχιστον για την χρονική περίοδο της αποθήκευσης των δεδομένων ούτε υπάρχει και καμιά καταληκτική ημερομηνία. Ε, αυτά είναι στοχευμένα. Και οφείλω να πω επίσης ότι εάν εξετάσουμε αυτή την στόχευση, ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής σήμερα πάνε προς μια καλύτερη κατεύθυνση από αυτή που πάμε εδώ στην Ευρώπη. Μιλάνε για targeting των μέτρων τους. Προσπαθούν να περιλάβουν τουλάχιστον κριτήρια στόχευσης. Λένε θέλουμε να περιλάβουμε, θέλουμε να συλλέξουμε τα δεδομένα ανθρώπων που η δραστηριότητά τους εμπεριέχει κάποιο ε, ρίσκο. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ζητάν κάποιο feedback από την πολιτική και ότι δεν βλέπουν καμία ανάγκη να συλλέγουν δεδομένα ε, συλλογής οποιονδήποτε προσώπων. Κοστίζουν πολλά λεφτά, χρόνο απασχόληση προσωπικού να αναλύσουν δεδομένα δηλαδή τα οποία είναι απολύτως άσχετα. Άρα χρειάζεται καλύτερη στόχευση και αυτό πρέπει να είναι η βασική ε, προσπάθειά μας. Αν θέλουμε να επιτύχουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ νομίζω μάλιστα ότι είναι πραγματικά σκανδαλώδες το ότι η Κομισιόν και το Συμβουλίο δεν έχουν αλλάξει την πρότασή τους μετά από τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άφησαν το περιεχόμενο της οδηγίας όπως είναι αγνοώντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι απολύτως παρανοϊκό. Και μάλιστα και αν σκεφτείτε ότι τα δεδομένα PNR είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα προσωπικά δεδομένα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αλλά ακόμα και αν σκέπτεστε έτσι, τότε εμεί στείλαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή έστειλε ξανά το σχέδιο συμφωνίας με τον Καναδά πάλι στο δικαστήριο για να ε, υπάρξει αναλογική μείωση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων τουλάχιστον το δικαστήριο να μπορέσει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ας αφήσουμε να απαντήσει τουλάχιστον πριν να προχωρήσουμε και ε, να εγκρίνουμε ταχύτατα κάτι το οποίο, ένα μέτρο ακόμα το οποίο θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Μιλώ λοιπόν για το θέμα αυτό, τη στόχευση. Και αν λύσουμε το πρόβλημα αυτό, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνένεση και τη κοινωνία, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και από πλευρά κοινωνία. Συνένεση την οποία δεν έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα με αυτή τη συνολική, την καθολική ε, ε συλλογή και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των επιβατών. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενοι στα θέματα αυτά, προσπαθώντας όμως να είμαι πάρα πολύ σύντομος ταυτόχρονα. Νομίζω το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε στη διάθεσή μας το Ευρωπαϊκό PNR. Βλέποντας όμως το πώς πηγαίνουν τα πράγματα σήμερα, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Το θέμα είναι ότι το υπάρχον σύστημα επιτρέπει σε όλο τον κόσμο να μετακινείται χωρίς ελέγχου στην Ευρώπη και αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία του εισηγητή που εργάστηκε εδώ και πολύ καιρό και πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέμα που προκαλεί πάρα πολλές αντιθέσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα με ψύχρεμο τρόπο για να επιλέξουμε ανάμεσα σε όλες αυτές τις εκατοντάδες τροπολογίες. Δεν έχουμε όμως ε, δυστυχώς τον χρόνο που απαιτείται και αυτό είναι ανησυχητικό. Στόχος μας είναι το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε μία κατάληξη των διαπραγματεύσεων που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να πάρουν τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την πρόληψη των τρομοκρατικών ενεργειών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ενδοκινοτικές πτήσεις, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι για το ποιόν των επιβατών οι οποίοι ε, μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σημασία όμως όλα αυτά να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν. Βλέπουμε τι έγινε από το 2011 και μετά και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και όλοι θα πρέπει να δεχθούμε την πρόταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιοι είναι οι ομιλητές στον κατάλογο. Η κυρία Ντονανό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τις ε, τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει και συνυπογράψει, θέλω να πω ότι στηρίζω τη συμπερίληψη ιδιωτικών πτήσεων και πτήσεων Charter στο μηχανισμό PNR, πολλές εκ των οποίων ε, πηγαίνουν είτε έρχονται από ε, ευαίσθητε περιοχέ. Έτσι θα είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα PNR αλλά και πιο δίκαιο σε σχέση με του παραδοσιακού αεροπορικού μεταφορεί. Επίση θα πρέπει να γίνει επιχειρησιακό περισσότερο το PNR, γι' αυτό και είμαι υπέρ τη κατάργηση ε, τη έννοια διακρατικό, όταν μιλάμε δηλαδή για τα σοβαρά δικήματα. Επίση, στη φάση τη έρευνα δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε εάν μία εκ πρώτη όψεω εθνική αξιόπινη πράξη θα μπορούσε να έχει διακρατικό χαρακτήρα. Το PNR το μόνο μπορεί να κάνει να βοηθήσει ε, να φανούν οι διακλαδώσεις ε, και οι συνένοχοι μπορεί να υπάρχουν ε, σε άλλες χώρες. Πρέπει να είναι αναλογικές οι διατάξεις. Εμείς έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες για να ενισχύσουμε τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ των ευαίσθητων δεδομένων που πρέπει να αποκλείονται, επιμένω να μην μπαίνει η έννοια φιλή θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές και δεν έχει κανένα νόημα κάτι τέτοιο, διότι όλοι στην ίδια φυλή ανήκουμε. Επίσης ε, και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ε, αν θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικό, επιχειρησιακό, αναλογικό και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα το σύστημα PNR, το ευρωπαϊκό σύστημα PNR θα έχει πραγματική προσθέμενη αξία για να αντιμετωπίσει τον κρανωμένο έγκλημα και την ε, τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκυγιόμ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, και η Σοφή, αλλά για ένα άλλο ε, θέμα, Αγουστίν και μένα με εξέπληξε αυτό. Και αν θέλετε να μας προκαλέσετε, τα καταφέρατε. Να πείτε στον Άξελ Βος να μην διαβάζει, να μην εμπιστεύεται τέλο πάντων τόσο πολύ τα γερμανικά δημοσιεύματα για την αποφυγή τρομοκρατικών επιθέσεων ε, και να ξέρετε ότι εμείς τις ε, αποφάσεις μας ε, τις παίρνουμε κατά αντιπαράσταση και αντιπαραβολή απόψεων και με άλλα θεσμικά όργανα ως θα καταθέσω τροπολογίες τέσσερα θέματα. Ενίσχυση ευρωπαϊκής διάστασης του συστήματος, άρα ότι μπορεί να εναρμονίσει, να έχει εναρμονιστικό αποτέλεσμα η οδηγία. Υπάρχει μια πρόταση η οποία διατηρεί την ε, κεντρική δομή και διαδικασία, αλλά θα πρέπει το σύστημα συνολικά να εποπτεύεται και να λειτουργεί με βάση κάποιες κοινέ βάσεις. Δεύτερο ε, είναι η βελτίωση των εγγύησεων με διάφορα υποσημεία τι στοιχεία πρέπει να δίνονται στους επιβάτες, τι πληροφορίες, ε, ότι πρέπει να βελτιωθεί επίσης ε, το σύστημα με τις ε, μονάδες πληροφόρησης των επιβατών, εγγύησης ό,τι αφορά τη μεταφορά δεδομένων που σε τρίτες χώρες και αξιολόγηση κινδύνων. Τρίτο, τι γίνεται με τα ευαίσθητα δεδομένα. Θα πρέπει να ενισχυθούμε τις εγγύσει ότι αυτή τη μεταβίβαση δεδομένων ευαίσθητων και θέλω κι εγώ στο παράρτημα να καταργηθεί η κατηγορία γενικές παρατηρήσεις. Τώρα, σε αυτή την πρόταση, όπως συχνά συμβαίνει άλλωστε, η επανεξέταση, η μεταγενέστερη επανεξέταση λέει ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε ποσοτικά σχεδόν κατά δεδομένα σε αυτή την αναθεώρηση. Εγώ νομίζω όμως ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να εστιάσει και σε ποιοτικά δεδομένα την αξιολόγησή της. Άρα μπορούμε να προσθέσουμε πιστεύω ορισμένα κριτήρια. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Um, what I wanted to do now... Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, στον εναπομένοντα χρόνο θα ήθελα να ζητήσω κάποιες απαντήσεις από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Δεν φαντάζομαι να μπορέσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της Σοφή η Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι εκπλήσεστε, Σοφή, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που θέλουμε τουλάχιστον να λάβουμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι κάποια απάντηση σε σχέση με την όλη συζήτηση. Πρώτα το Συμβούλιο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση είναι ότι το θέμα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σωστή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οδηγεί στη σημερινή συζήτηση και στην πρόταση του εισηγητή. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ψηφοφορία το ταχύτερο δυνατόν. Το Συμβούλιο παραμένει αποσιωμένο στην προσπάθεια έβρεσης μιας συμφωνίας. Όπως ακούστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στις διοργανικές επαφές. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρξει ένα ισχυρό πρόγραμμα PNR ευρωπαϊκό και η συνεισφορά του Κοινοβουλίου θα είναι πολύτιμη. Η Προεδρία συνειδητοποιεί επίσης τη μεγάλη σημασία που έχει και το πακέτο προστασίας και θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην λήψη των απαιτούμενων νομικών μέτρων Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να περάσουμε σε λεπτομέρειες. Έχουμε εκτιμήσει ήδη έχουμε δηλώσει την εκτίμησή, σας, την εκτίμησή μας στην προσπάθειά σας να υπενθυμίσω προς την κυρία Ιντβελτ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει με επιστολή στο ψήφισμα της 11ης Φεβρουαρίου απεστάλει στο Κοινοβούλιο στις 11 ακριβώς Φεβρουαρίου και εντοπίζουμε στην απάντησή μας αυτή στοιχεία τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι απάντηση. Τώρα για την επιστολή της κυρίας Σίντβελτ τον μήνα Μάρτιο θα τύχει απάντηση στο ταχύτερο δυνατόν. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος θα σας στείλει μια επιστολή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Είχατε θέσει συγκεκριμένες λεπτομερείς ερωτήσεις Ενθυμίστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οργανώσει δύο συναντήσεις, τη μία μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά ε, επίσης την άλλη από δική της πρωτοβουλία. Νομίζω ότι έτσι δόθηκε η ευκαιρία και σε κοινοβουλευτικούς να πάρουν απαντήσεις από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, προφορικά. Νομίζω οι προφορικές αυτές απαντήσεις καλύπτουν πολλές από τις ανησυχίες ε, που περιλαμβάνονται στην επιστολή. Ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών ε, δεν δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπεράσει τα μέσα τα οποία τα κράτη-μέλη μας έχουν δώσει. Στα πλαίσια της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων υπήρξαν εθνικοί εμπειρογνώμονες όπως είπα αλλά και πολλοί κοινοβουλευτικοί. Εμείς μεταφέρουμε απλά τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι εθνικοί εμπειρογνώμονοι και πολλοί ευρωβουλευτές ε, ε, άκουσαν τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων. Τώρα για την ε, αναλογικότητα και την αναγκαιότητα. Το θέμα της αναλογικότητας συνδέεται με τις ρήτρες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή λειτουργήσει το PNR έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στα προσωπικά δικαιώματα, στα θεμελιώδη δικαιώματα και αν κάτι τέτοιο συμβεί να είναι απολύτως τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα τώρα. Όπως έχει επανειλημμένα υποθεί και στα πλαίσια της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων, το σύστημα PNR έχει σαν αποκλειστικό στόχο τον εντοπισμό των υπόπτων και την διεξαγωγή μιας έρευνας ή μιας ανάκρισης και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά με τα άλλα στοιχεία και τις άλλες μεθόδους που μετέρχονται οι δυνάμεις ασφαλείας. Είναι μερικές φορές δύσκολο να διακρίνει τις διαφοροποιήσεις όπου κάποια ευρήματα PNR οδήγησαν στην πρόοδο κάποιων γενικότερων ερευνών και που ε, οδήγησαν στην αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών ή πράξεων της διεθνούς εγκληματικής δραστηριότητας. Όπως είπα, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος θα σας αποστείλει την επιστολή του μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είδα, Σόφη, ότι ζητάς πάλι το λόγο. Επί τη βάση λοιπόν της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας ακούσαμε ότι θα πάρετε μια επιστολή από τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά θα σου δώσω το λόγο, αλλά παρακαλώ να είσαι πάρα πολύ σύντομη. Μου χρειάζεται κανένα λεπτό Περιμένω, αγαπητέ κύριε, συγκεκριμένη απάντηση στα συγκεκριμένα με ερωτήματα. Εργάζομαι για το θέμα αυτό 11 χρόνια. Ποτέ δεν έχω λάβει μια συγκεκριμένη απάντηση. Αν μου δώσετε μια απάντηση που να λέει η γη είναι στρογγυλή, Εντάξει, σωστό είναι και αυτό, αλλά δεν απαντάει στα ερωτήματά μου. Αν δεν έχουμε απαντήσει στα ερωτήματά μα, δεν ε, θεωρώ ότι ε, ισχύει και η δέσμευση, τουλάχιστον η δική μου δέσμευση, να εργαστώ για αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι και προσιλωμένοι, άρα και εσεί πρέπει να το αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα το θέμα και να μου δώσετε μια σοβαρή απάντηση. Αλλιώ δεν, δεν δουλεύουμε. Διευκρινίζω αυτό που είπα για τη γη και το Γαλιλαίο. Θα σου στείλω μια επιστολή σχετικά. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους έλαβαν το λόγο. Ως εισηγητής ε, ε, θα είχα το δικαίωμα να συνοψίσω. Άκουσα τις απόψεις όμως των συναδέλφων. Αυτό ήταν το σημαντικό και επίσης καλό ήταν που ακούσαμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να πω λοιπόν και να ξεκαθαρίσω σε όλους όσους μίλησαν σήμερα ότι θα συνεχίσω και μέχρι στιγμής αυτό έκανα άλλωστε, θα συνεχίσω να κάνω πάντο δυνατό για να συντονίζω τη συζήτηση και στο μέτρο του δυνατό να προτείνω συμβιβασμού που να βρουν όλο και όσο να δω περισσότερου συναδέλφου ικανοποιημένου. Βέβαια, υπάρχει ανησυχία και με ανησυχεί και εμένα ε, για το χρονοδιάγραμμα. Τρία μισή χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα. Μπορεί και να μην είναι ρεκόρ στο Κοινοβούλιο, αλλά κοντεύουμε να το σπάσουμε το ρεκόρ παρόλα αυτά. Και θέλω να πω ότι Νομίζω ότι πρόοδο σημειώνουμε. Μπορεί να μην είναι τόσο ταχεία όσο θα ήθελαν ορισμένοι, όμως προσωπική μου άποψη ηγητή είναι ότι έχω καθήκον να ακούσω τις διάφορες απόψεις και αν μπορώ να καταλήξω σε κάποιες συμφωνίες. Αυτή θα συνεχίσει να είναι η προσπάθειά μου μέσα στο χρονοδιάγραμμα της, ε, που έθεσε η Ολομέλεια και αν μπορώ να έχω τις υποστήριξεις όλων των ομάδων ε, και των μεγάλων και των υπόλοιπων, για να το πετύχω αυτό θα είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μεσικής Διάταξης. Ευχαριστώ. Which is uh, mandate, it's, point it's mandate for opening negotiations for an... E και αυτό είναι το σημείο 8, δηλαδή εντολή για την άνοιξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία PNR Α, PNR, κάτι τελείω διαφορετικό. Μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού. Λοιπόν, μα ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ότι από τον Νοέμβριο του 2012 έχει το Μεξικό λομοθεσία για το PNR και απαιτεί από όλου τι ευρωπαϊκέ εταιρείε που έχουν πτήσει από και προ Μεξικό να διαβιβάσουν στοιχεία PNR. Και παρακαλώ να σταματήσουν οι συζητήσει. Λοιπόν, το Μεξικό ανέφερε ότι εταιρείε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι μόνε που δεν δίνουν στοιχεία PNR στι μεξικανικέ αρχέ. Όμω η μεξικανική νομοθεσία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ για τι ε, αεροπορικέ εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Κομισιόν ζήτησε από το Μεξικό να αναβάλει την επιβολή προστήμων ε, για διάφορε περιπτώσει. Οι αρμόδιε αρχέ του Μεξικού κατέστησαν σαφέ νωρίτερα φέτο ότι η τελική ημερομηνία, η τελική προθεσμία για την μεταφορά στοιχείων PNR είναι η 1η Απριλίου του 2015. Ο Επίτροπο Αβραμόπουλο, μιλώντα στην Ολομέλη τον Απρίλιο δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές του Μεξικού συμφώνησαν για αναβολή ε, της ε, προθεσμίας μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεσμευτεί να ξεκινήσει επίσημα διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Κομισιόν λοιπόν ζητά εντολή από το Συμβούλιο για επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων και μια συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. Ωστόσο, ο Επίτροπος δήλωσε επίσης ότι μια συμφωνία PNR με το Μεξικό δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί προτού γνωμοποιηθεί γνωμοδοτήσει το δικαστήριο για το σχέδιο συμφωνίας PNR με τον Καναδά και ότι γνωρίζουν ότι περί αυτού πρόκειται οι μεξικανικές αρχές. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις, όλοι μας, όλοι μας θα ήθελαμε κάποιες διευκρινήσεις, θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ενημερώσει επί του θέματος, να μας πει πως έχει κατάσταση. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας ζητάτε να σας ενημερώσουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία για να σας επιβεβαιώσω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και ζητά από το Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Μεξικό για το PNR. Ήμασταν δεσμευμένοι στην εξέβρεση μιας νέας λύσης στο ζήτημα της διαβίβασης δεδομένων PNR ε, για πτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Μεξικό έχει ε, τη σχετική νομοθεσία από τον Νοέμβριο του 2012 και αυτή η νομοθεσία απαιτεί όλες τις αεροπορικές εταιρείες ε, που κάνουν τις από και προς το Μεξικό να, μεταφέρουν, να μεταβιβάζουν τα δεδομένα PNR. Από τότε λοιπόν και μετά όσοι φορείς, όσοι μεταφορείς δεν μεταφέρουν, δεν μεταβιβάζουν αυτά τα στοιχεία μπορεί να τους επιβληθούν κυρώσεις. Όμως ό,τι αφορά της πτήσης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία γιατί ζήτησε αναβολή η Κομισιόν από το Μεξικό την επιβολή προστήμων σε διάφορες ε, περιπτώσεις. Ε, καταφέραμε να έχουμε αυτή την αναβολή σε διάφορες περιπτώσεις. Ε, τελευταία το Μεξικό κατέστησε σαφές ότι η τελευταία ημερομηνία για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων είναι η 1η Απριλίου και ζήτησε να γίνει κάθε ε, προσπάθεια για να μην επιβληθούν οι κυρώσει στις αεροπορικές ε, εταιρείε. Ο Επίτροπος ε, Αβραμόπλος είναι σε συνεχή επαφή με τις μεξικανικές αρχές του τελευταίους μήνες. Και περί τα τέλη Μαρτίου συγκεκριμένα ζήτησε και την αναβολή της προθεσμίας. Ενημέρωση Κομισιόν το Μεξικό ότι προτίθεται να προτείνει στο Σώμα των Επιτρόπων να ζητήσει εντολή από το Συμβούλιο. Όπω γνωρίζετε, αυτό οδήγησε σε αναβολή τη προθεσμία από το Μεξικό και η νέα προθεσμία είναι η 1η Ιουλίου. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια σύσταση προ το Συμβούλιο για επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού. Η πρόταση να ζητηθεί εντολή για έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε δεκτή θετικά από το, Κομισιο και όπως, από το Μεξικό και όπω είπα, ε, ζητούμε και την αναβολή των προστήμων, της των προστήμων. Είναι ε, δύσκολο να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό ε, πρόκειται για την ίδια εντολή με αυτή που έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις για διαπραγματεύσει συμφωνίας PNR. Έχουμε και την ανακοίνωση του 2010 που αποτελεί μια καθοδήγηση για εμάς, όπως επίσης και η διατάξει του ψηφίσματο του Κοινοβουλίου πάλι του 2010 και έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για την οδηγία περί διατήρησης δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη, σαφώς, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις οι οποίες θα λάβουν υπόψη την άποψη ή μάλλον καλύτερα την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Είπατε κι εσείς κύριε Πρόεδρε ότι οι μεξικανικές αρχές έχουν κατανοήσει το θέμα, ότι δηλαδή αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν και δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν προτού έχει εκδώσει την ε, γνωμοδότησή του το δικαστήριο σε σχέση με την Συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε άλλη χώρα ζητήσει ε, κάποια δεδομένα PNR από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος τη σύσταση ολοκληρώνει το έργο του και αναμένουμε ότι θα έχουμε απόφαση σύντομα με την προπόθεση ότι το Συμβούλιο θα μας δώσει την εντολή, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Προβλέπεται αυτό να γίνει περί τις αρχές Ιουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να έρχεται στη ΛΥΜΠΕ και να σας ενημερώνει για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όσο αυτές διαρκούν, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε μας το ζητήσετε. Σας ευχαριστώ. Thank um, got... Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις ομιλητές. Η κυρία Ίντεβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή της, για την παρουσίαση. Χαίρομαι που προχωρούν πλέον τα πράγματα. Διερωτώ με τι έχει εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσα χρόνια να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους Μεξικανούς. Μας κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι πηγαίνουμε αργά στα πλαίσια του PNR. Εγώ θέτω το θέμα με τις τρίτες χώρες εδώ και τρία χρόνια. Έχω τρεις σελίδε εγώ με τις επιστολές και τις ερωτήσεις που έθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο με το Μεξικό, για το Μεξικό, αλλά η Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Νότιο Αφρική, Μαλαισία κτλ. Οι Ιάπωνες είπαν ότι δεν θα περιμένουμε, εμείς θα ξεκινήσουμε μονομερό στη συλλογή Πιονάρ η ΙΑΤΑ λέει στους αερομεταφορείς να υπακούσουν στην Ιαπωνική νομοθεσία που παραβιάζει όμως τον κοινοτικό νόμο. Συνεπώς λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω σε καμία περίπτωση τον λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κινείται. Τι σας εμποδίζει γιατί δεν συζητάτε με τους ε, Ιάπωνες ή Νοτιοκορεάτες παρακαλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθούν. Και η συμφωνία αυτή είναι και προς το δικό μας συμφέρον, όχι μόνο προς το δικό τους. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Χαίρομαι που κατεκινείτε για το Μεξικό. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά τι θα κάνετε με τις άλλες χώρες. Ε, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά. Δεν είναι όλες οι χώρες αυτές φιλικές δημοκρατίες ε, με νόμους αντίστοιχους με τους δικούς μας. Γι' αυτό λοιπόν τι σας εμποδίζει, τι θα κάνετε με τις χώρες αυτές, πότε επιτέλους θα ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις και για πόσο καιρό τα δεδομένα μας θα πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες χωρίς η μορφή προστασίας. Σας... Ο πρόεδρος κ. να διευκρινίσω κάτι, Σοφή. Το 1850 ένας έγραψε ένα βιβλίο και εκεί ορισμένοι υποστηρίζουν και υπάρχει ακόμα μια τέτοια ε, ε, ένωση στην Μεγάλη Βρετανία ότι η ε, γη είναι επίπεδη. Ο κύριος Ντεμέρα, ευχαριστώ πολύ. Ακούω με μεγάλο σεβασμό τους συναδέλφους και διδάσκομαι από αυτούς. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να με ακούν και οι συναδελφοί μου με σεβασμό και να καταλαβαίνουν τη διαφορά. Άλλο να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο και άλλο να λέω ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση είπε ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος είπε. Δεν αποσύρω ούτε ένα κόμμα από την προηγούμενη παρέμβασή μου, αλλά επαναλαμβάνω με κάθε σεβασμό προς όλους τους συναδέλφους. Τώρα, δεν θέλω να ασκήσω κριτική, αλλά κάπως να θέσω που αμφισβήτηση αυτό που είπε η Κομισιόν. Λοιπόν, είπατε απαγόρευση ε, ή μάλλον ε, μία περίοδος χάριτος, αν θέλετε, που θα λήξει 1η Ιουλίου. Ποια είναι η διαδικασία. Έχουμε το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λέει ότι κατόπιν ετήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για διαπραγματευτική εντολή, όπως και μας είπε η Κομισιόν, το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο με απόφασή του δίνει ή δεν δίνει αυτή τη διαπραγματευτική εντολή. Η προθεσμία που έχουμε μπροστά μας όπως φαίνεται είναι, και να προσέξετε παρακαλώ τι σας λέω. 9 Ιουνίου το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε επίπεδο κορεπέρ. Με την ελπίδα, και παραλαμβάνω με την ελπίδα να ψηφιστεί από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στις 23 Ιουνίου. Άρα, 9 Ιουνίου, 23 Ιουνίου. Υπάρχει όμως και κάτι που με ανησυχεί. Γι' αυτό και είπα ότι υπογραμμίζω τη λέξη ελπίδα με την ελπίδα. Διότι υπάρχουν αμφιβολίες εντό Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη νομική βάση που πρέπει να εφαρμοστεί. Έχουμε τα πρωτόκολλα 21 και 22 που αναφέρονται στο Ενωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Για τη δική μου πολιτική ομάδα και για τη χώρα μου όμως ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, είναι προτεραιότητα για εμάς. Θα ήθελα λοιπόν, εάν θεωρείτε ότι αυτή η πολύ σύντομη ε, χρονική πεσμία είναι αρκετή για να ε, διασκεδαστούν οι αμφιβολίες ό,τι αφορά τη νομική βάση. Δεν ξέρω αν σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πολύ αμφιβάλλω. για να πάρει και η Κομισιόν τελικά την απόφαση, δηλαδή τη διαπραγματευτική εντολή για την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων με το Μεξικό. Ακούστε τι θα πω, ε, το είπα ε, και στην Ολομέλεια. Ένα στοιχείο. Το πρόστιμο 30.000 ευρώ αναπτύσσει είναι πάρα πολύ ψηλό πρόστιμο. Η Ιμπέρια, η εταιρεία της χώρας μου, έχει λάβει την προειδοποίηση ότι το Μεξικό θα εφαρμόζει πρόστιμα ακόμη και για έξι επιβάτες αναπτύσσει. Για την Ιμπέρια που έχει δύο καθημερινέ πτήσει και 7 μέρες την εβδομάδα, αυτό σημαίνει πρόστιμα των 320.000 το μήνα, 16 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα με ανησυχεί το ότι ενημερώνει η Κομισιόν για πράγματα που είναι αόριστα και ασαφή. Εγώ θέλω να μας πει πραγματικά η Κομισιόν αν η νομική βάση ισχύει ή δεν ισχύει και αν θα υπάρξουν ή όχι προβλήματα εντό του Συμβουλίου, γιατί είναι πολύ λίγες ημέρε που έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Sippel. Thank you. Ευχαριστώ Σίπελ. Εγώ επιθυμώ να προσεγγίσω το θέμα διαφορετικά και θέτω το ερώτημα γιατί διαπραγματευόμαστε καν με το Μεξικό για αυτό το σύστημα PNR έτσι, διότι το Μεξικό αποφάσισε και θέλει τα δικά μας προσωπικά δεδομένα. Άρα, δηλαδή, εν τέλει, διαπραγματευόμαστε με οποιονδήποτε, δηλαδή με την Κορέα, με τη Ρωσία, όποιοι θέλουν να τους δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Αν δεν κάνουμε συμφωνία, τότε λένε ορισμένοι, μα ή άλλως θα τα πάρουν τα δεδομένα και μάλιστα σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δικαίωμα. Γιατί διότι υπάρχουν κάποια οικονομικά συμφέροντα τα οποία είναι ισχυρότερα από το ερώτημα τι γίνεται στο Μεξικό, στη Βόρεια Κορέα ή στη Ρωσία, δεν ξέρω πού αλλού, τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών μας. Εκεί νομίζω πρέπει να στοχεύσουμε. Εκεί πρέπει να συζητήσουμε. Όχι αν υπάρχει συμφωνία ή όχι, αλλά το τι γίνεται πραγματικά. Και αν θέλουμε και πραγματικά να πούμε κάποια στιγμή στους πολίτες τι γίνεται και αν φέρνουμε κάποια αντίσταση ή όχι όταν διαδίδονται περαιτέρω τα δεδομένα αυτά. Εκεί πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις. Εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη όταν βλέπω τις ειδήσει από το Μεξικό για το εάν αυτό το Μεξικό είναι πραγματικά μια χώρα που μπορεί να επαφίεται κανείς ότι υπάρχει μια δημοκρατική αντίληψη σε ό,τι αφορά την δράση των αστυνομικών δυνάμεων και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και πέραν του ερωτήματος τώρα εάν η διαδικασία είναι καλή ή κακή. Ευχαριστώ εξάλλου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δηλώνει διατεθειμένη να επανέλθει να μας ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως οποιαδήποτε άλλη στάση θεωρώ ότι θα ήταν απαράδεκτη, να μην έρθει δηλαδή. Ευχαριστώ λοιπόν που λέει κάτι το αυτονόητο. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω, εφόσον αποδίδουμε αξία στις δημοκρατίες που συναπαρτίζουν την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, που φροντίζουν για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της προσωπικής σφαίρας. Έχω κάποια φορά την εντύπωση ότι όλα αυτά τα πράγματα ναι μεν ηχούν ωραία, αλλά στην πράξη αν κάποιοι οικονομικοί λόγοι το υπαγορεύουν, είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε τις αξίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννα Άλμπρεχτ. Στα Αγγλικά, ο κύριος Άλμπρεχτ. Εγώ ευχαρίστω να λάβω το λόγο μετά από αυτά που λέχθηκαν για τα αρχεία ονομάτων επιβατών PNR που τα έχουμε συμφωνήσει με Αυστραλία, Ενωμένε Πολιτείε, Καναδά και βέβαια και σε παραβίαση της απόφασης του δικαστηρίου είναι καθαρό ότι το να στέλνουμε όγκους ολόκληρους ε, δεδομένων επιβατών ε, έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του δικαστηρίου για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του χάρτη. Άρα, αντί να εγκρίνουμε παραπάνω τέτοιες συμφωνίες, καλύτερα να θεωρήσουμε τις υφιστάμενες. Και χαίρομαι που το, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να διαβιβάσει τη συμφωνία αυτή στο δικαστήριο για να την εξετάσει αν δηλαδή είναι σύνομη με την κείμενη νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μου φαίνεται λίγο παράξενο να συζητούμε μέσα στα πλαίσια της οδηγίας PNR εάν θα πρέπει να κοινοποιούνται και μεταξύ των χωρών μελών όλα αυτά τα PNR και να λέμε όχι, αλλά να τα διαβάζουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου που επιβάλλει κυρώσεις, εάν ή θα απειλεί θα μας επιβάλλει κυρώσεις, αν δεν το πράξουμε. Αυτό μου φαίνεται λίγο παράξενο. Να πούμε καθαρά λοιπόν ότι δεν είναι τρόπος αυτός, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε να το περιορίσουμε, θέλουμε να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας με τους εταίρους μας εφόσον και αυτοί έχουν κράτη ε, βασισμένα στην ισχύ του δικαίου κτλ. Αυτά. Ε, γιατί έχω μεγάλη εμφιβολία για το κράτος δικαίου του Μεξικού. Ευχαριστώ. Κύριε Χοπ, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επανέλθει, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στα εκλεκτά μέλη. Για την κυρία Ιντβέλτ, όπως είπα στην αρχική μου παρουσίαση, η νομοθεσία του Μεξικού τέθηκε σε εφαρμογή από τα τέλη του 2012. Μέχρι τότε δεν είχαμε κάποια επαφή και δυνατότητα επαφής στα πλαίσια του τεχνικού διαλόγου για να κατανοήσουμε τις ρυθμίσεις τους. Τους υποβάλαμε ερωτηματολόγιο για να συλλέξουμε πληροφορίες, να δούμε ακριβώς τι είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν και αυτό κάναμε και παλιότερα. Αυτό απαιτεί χρόνο. Ε, επισκεφθήκαμε το Μεξικό και εγώ προσωπικά πήγα εκεί και οι αρχές του Μεξικού έχουν έρθει εδώ. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο έτσι ώστε να συλλεγούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και να έχουμε μια κατάλληλη εντολή. Αυτά σχετικά με τον χρονισμό. Για τις υπόλοιπες χώρες, μια οριζόντια αντιμετώπιση είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε και αυτό το λέει και στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα ασφαλείας. Εμείς έχουμε προτείνει στο Συμβούλιο ε, μια συμφωνία πρότυπο. Πάντως θα πρέπει να περιμένουμε, όπως φαντάζεστε, από την ε, γνωμοδότηση του ECJ για τον Καναδά, να ξέρουμε τι θέλει το δικαστήριο δηλαδή, πριν προχωρήσουμε στην καθιέρωση των κριτηρίων τα οποία μπορούμε να επιβάλλουμε σε τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν πρέπει να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα. Ε, λέτε ότι η συμφωνία είναι επίσης προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς το συμφέρον της Ένωσης, θα είναι και νομική υποχρέωση. Το 25.2 της οδηγίας του 95 υποχρεώνει στα πλαίσια μιας νομικής ε, διεθνούς συμφωνίας να καλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν υπάρξει μια διεθνή συμφωνία, θεωρητικά δεν μπορεί να γίνεται και είναι παράνομη η ανταλλαγή στοιχείων. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε τώρα για τον κύριο Διαστεμέρα. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στο άρθρο 218. Αυτή ήταν η νομική βάση. Και γι' αυτό ακριβώς ε, ε, στείλαμε την μπάλα στο Συμβούλιο και τώρα πρέπει να απαντήσει το Συμβούλιο και δεν θα πάρω εγώ το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Συνειδητοποιούμε τις συγκεκριμένες συνέπειες που θα είχε η καθυστερημένη αποδοχή για τον κίνδυνο μεταφοράς προσωπικών δεδομένων χωρίς μια διεθνή συμφωνία. Τέλος, για την κυρία Τσίπελ. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι οι χώρες είναι ε, κυρίαρχες. Θέλει να εφαρμόσει την εθνική του νομοθεσία. Είναι στρατηγικός εταίρος βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό απαιτείται μια συμφωνία έτσι ώστε να μην υπάρχει μη συντονισμένη αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη τη απουσία συμφωνίας. Ευχαριστώ. Είπατε ότι δεν θα πάρετε τον λόγο για το Συμβούλιο συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. να επιβεβαιώσω ότι τα κράτη-μέλη ζητούν να υπάρξει μια συγκεκριμένη εντολή εδώ και αρκετό καιρό. έτσι ώστε να αναβληθούν πιθανές κυρώσεις από πλευράς του Μεξικού. Ο χρόνος πιέζει όπως είπαμε και γι' αυτό εμείς Είμαστε υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να περάσει η πρόταση από τα προπαρασκευαστικά στάδια της διαδικασίας του Συμβουλίου. Δεν εργούμε. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα στην υιοθέτηση της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να υπάρξει μία απόφαση του Συμβουλίου πριν από το τέλος του μηνός Ιουνίου. Και ελπίζουμε ότι αντίστοιχες προθεσμίες θα ακολουθήσει και η μεξικανική πλευρά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους ήσαν παρόντες. Έτσι κλείνει η συζήτησή μας για σήμερα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί στις 3 το μεσημέρι. Διακόπτουμε.